Okay, I think we should get started. Welcome everybody. We have... Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Έχουμε αρκετά φορτωμένη μέρη σε διάταξη για σήμερα και θα πρέπει να ξεκινήσουμε εάν δεν υπάρχουν σχόλια μπορούμε να την νομίζω όπως συνήθως ε, η σημερινή συνεδρίαση μεταδίδεται μέσω web streaming. Υπάρχει δερμηνία σε όλες τις γλώσσες. Έχουν σταλεί τα πρακτικά της συνάγκη των συντονιστών στις 17 Οκτωβρίου. Μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα στα πρακτικά. 17 Οκτωβρίου επαναλαμβάνω είναι η συνεδρίαση. Δεν υπάρχουν σχόλια. Πολύ ωραία. Περνάμε στο σημείο 4 και εδώ με μεγάλη χαρά θα καλωσορίσω την κυρία Πάουλα Πίνιο, η οποία αυτή τη στιγμή είναι διευθυντή ε, στη Γενική Διεύθυνση Ενέργεια ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μα παρουσιάσει την ενεργειακή κοινότητα και την αναθεώρηση ε, τη συνθήκης που θεσπίζει, που δημιουργεί την ενεργειακή κοινότητα. Όπω ξέρετε πρόκειται μια διεθνή οργάνωση όπου συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι γείτονέ τη για να έχουμε ε, ένα ενοποιημένο, ένα, μια ενιαία ενεργειακή αγορά πανευρωπαϊκή. Τον Οκτώβριο του 2005 είχε υπογραφεί αρχικά αυτή η συνθήκη στην Αθήνα και εφαρμόζεται από το 2006. Ο βασικός στόχος της ενεργειακής κοινότητας είναι να επεκτείνει τους κανόνες της, εσωτερική της εσωτερικής αγοράς της ενεργειακής, τους κανόνες και τις αρχές στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, στη Μαύρη Θάλασσα, επί τη βάση μιας δεσμευτικ, ενός δεσμευτικ, νομικός δεσμευτικού πλαισίου. Ε, κυρία Πίνιο, σας δίνω το λόγο. Έχουμε μία ώρα για την όλη συζήτηση. Ε, έχετε το λόγο. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ και μπορώ να μιλήσω για την ενεργειακή κοινότητα. Είχα ε, την πρώτη συζήτηση ε, εδώ, έχω την πρώτη συζήτηση εδώ ε, σε αυτή τη νέα θητεία του Κοινοβουλίου. Η ενεργική κοινότητα όντως φέρνει μαζί, φέρνει κοντά την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κρατημέλη της και εννέα συμβαλόμενα μέρη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, Αλβανία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Βόρεια Μακεδονία, Κόσοβο, Μαυροβούνιο και Σερβία. Επίσης, ε, τρεις χώρες της Ανατολικής ε, Γειτονίας, Γεωργία, Ουκρανία, Μολδαβία. Δημιουργήθηκε ε, μέσω της συνθήκης του 2005 για την ενεργή κοινότητα που τέθηκε σε συνθήκη το 2006. Ε, πρόκειται για ένα εργαλείο κλειδί της ε, εξωτερικής πολιτικής ε, της Ένωσης. Ο βασικός στόχος της ενεργικής κοινότητας είναι να δημιουργήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο για μια ενοποιημένη ενεργειακή αγορά, περιφερειακή ενεργειακή αγορά, μεταξύ των συμβαλωμένων μερών δηλαδή, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι μια ενεργειακή ενιαία αγορά δεν σταματάει στα σύνορα ε, της Ένωσης. Η ροή τη ηλεκτρικής ενέργεια ε, πάει και παραπέρα. Έχουμε κάτι συμφέρον λοιπόν να επεκτείνουμε του κανόνε μα εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπογράφοντα αυτή τη συνθήκη, τα συμβαλόμενα μέρη έχουν δεσμευθεί για να εφαρμόσουν σημαντικέ νομοθεσίε στον τομέα τη ενέργεια εντό συγκεκριμένου χρονικού διαστήματο. Ε, υπάρχει μια διαδικασία επίλυση διαφορών. Αυτό εξασφαλίζει την εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουν αναλυφθεί. Η ενεργειακή κοινότητα λοιπόν είναι ένα σημαντικό καταλήτη για την ανάπτυξη τη ενέργεια στην περιοχή και αυτό μπορεί να έχει και επιπτώσεις σε άλλους τομείς πολιτικής. Πέρα από τον στόχο της δημιουργία ενός σταθερού ρυθμιστικού πλαισίου για την αγορά που να ε, προσελκύει τις επενδύσεις και να ενισχύει ε, την ασφάλεια των εφοδιασμού πρέπει να βελτιωθεί και η περιβαλλοντική κατάσταση σε ό,τι αφορά την ενεργεια, τον ενεργειακό εφοδιασμό, να ενισχύσει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργεια και τη αποδοτική χρήση ενέργεια και ε, να αναπτυχθεί ο ανταγωνισμό σε περιφερειακό επίπεδο και να εκμεταλλευτούμε τι οικονομίε κλίμακα. Ε, σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση τη ενεργειακή κοινότητα, το βασικό όργανο ε, που παίρνει τι αποφάσει είναι το Υπουργικό Συμβούλιο, που συνέρχεται μια φορά το χρόνο στην χώρα που, ε, αναλαμβάνει την Προεδρία τη Ενεργειακή Κοινότητα. Αυτή τη στιγμή είναι η Μολδαβία η χώρα αυτή και θα επανέλθω από αυτού στη συνέχεια, μια και η ενεργεια, το Υπουργικό Συμβούλιο θα συνέλθει στι 15 Δεκεμβρίου στο Τσιτσινάου. Υπάρχει μια ομάδα που, που συνεδριάζει τέσσερι φορέ το χρόνο και που προετοιμάζει την Υπουργική Σύνοδο. Υπάρχει η Γραμματεία τη Αλληλεγγύη Κοινότητα που είναι το εφαρμοστικό όργανο, το εκτελεστικό όργανο, συγγνώμη, και το Ρυθμιστικό Συμβούλιο που είναι ένα ανεξάρτητο ε, σώμα ρυθμιστικών αρχών. Ε, και συμμετέχει εκεί και η ΕΣΑ, το όργανο Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών. Υπάρχει ένα θέμα ε, βελτιωμένης εφαρμογής ε, του κεκτημένου και υπάρχει εδώ μια κοινοβουλευτική διάσταση ε, στην ενεργειακή κοινότητα. Υπάρχει μια ολομέλεια η οποία ε, συνέρχεται δύο φορές το χρόνο υπό την Προεδρία του Κοινοβουλίου της χώρας που έχει αναλάβει την Προεδρία και του Υπουργικού Συμβουλίου. Η επόμενη συνάντηση θα λάβει χώρα ε, στις 12 Δεκεμβρίου φέτος. Αυτό αυτή η κοινοβουλευτική ολομέλεια ε, αποτελείται από δύο κοινοβουλευτικού εκπροσώπου από την ΚΑΠ, το καθένα από τα συμβαλόμενα μέρη, και εκπροσώπους βεβαίως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, αυτή η Ολομέλεια εκφράζει άποψη για όλα τα ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο της ε, συνθήκης ε, με ψηφίσματα με την εξαίρεση της επίλυση διαφορών. Μπορούν επίσης να θέσουν ερωτήσεις στα όργανα της ενεργειακής κοινότητας. Αυτά σε ό,τι αφορά το ευρύτερο πλαίσιο, σε ό,τι αφορά τώρα τα βασικά ζητήματα τα οποία μας απασχολούν αυτή τη στιγμή στην ενεργειακή κοινότητα, ε, θα αναφερθώ σε δύο σημεία κυρίως. Πρώτον, η μεταρρύθμιση της ενεργειακής κοινότητας και της σχετικής συνθήκης και οι τροποποιήσεις ε, που θέλουμε να επιφέρουμε εκεί και οι στόχοι του 2030 για το κλίμα. Σε σχέση με την ε, συνθήκη της ενεργειακής κοινότητας, η συνθήκη περνάει αυτή τη στιγμή από μια διαδικασία μεταρρύθμισης με σκοπό η ενεργειακή κοινότητα να γίνει πιο αποτελεσματική και να προσαρμοστεί σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Οι συζητήσεις για την τροποποίηση της συνθήκης ξεκίνησαν το 2016 μετά την έκθεση για την μετάδοση της ενεργής κοινότητας της μόνιμης ομάδας ψηλού επίπεδου του 2014 ε, τη οποία προέδρευσε ο κύριος Μπούζεκ, τον οποίο γνωρίζετε καλά. Μετά από αυτή την ε, έκθεση της ομάδας ψηλού επίπεδου, το 2017-2018 το Συμβούλιο ενέκρινε ε, διαπραγματευτικές εντολές για την τροποποίηση της συνθήκης ενεργειακής κοινότητας. τα βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης και της διαπραγμάτευσης είναι μια ιδιαίτερη αναφορά στην κλιματική πολιτική και των δεσμεύσεων που αναλάβαμε στα πλαίσια της Συμφωνίας των Παρισίων, η ενίσχυση της του μηχανισμού εφαρμογής μέσω ενός συστήματος κυρώσεων, στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με την συνθήκη της ενεργειακής κοινότητας και διαφάνεια σε ό,τι αφορά τον τομέα των κρατικών ενισχύσεων. Επίσης υπάρχει περαιτέρω ε, ολοκλήρωση της ενεργειακής ε, αγοράς ε, μέσω αμοιβαίων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και της, των συμβαλόμενων μερών της ενεργειακής κοινότητας. Πρόκειται για έναν μηχανισμό αμοιβαιότητας, έτσι ονομάζεται. Η όλη μεταρρύθμιση της συνθήκης της ενεργειακής κοινότητας έχει ξεκινήσει από εσά, κυρία Μπούζεκ, και την έκθεσή σας. Ε, πριν από μερικά χρόνια και χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ σήμερα και συζητούμε τη συνέχεια που θα δώσει αυτή την έκθεση. Τώρα, πού βρισκόμαστε στις διαπραγματεύσεις της μεταρρυθμιστής συνθήκης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζει ότι θα υπάρξει ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων αυτών εν ώψη της Υπουργικής Συνόδου του Δεκεμβρίου φέτος έτσι ώστε να ξεκινήσει το κείμενο αυτό στη Μολδαβία σύμφωνα με τη συνθήκη η έγκριση από το Συμβούλιο αλλά και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτείται στη συνέχεια πριν εγκριθεί το τελικό κείμενο. Έτσι λοιπόν η Επιτροπή Ήτρε θα εξετάσει το ζήτημα αυτό εφόσον ολοκληρώσουμε το Δεκέμβριο με το κείμενο αυτό στην Υπουργική Σύνοδο και ε, βεβαίως αναμένουμε συνεργασία μαζί σας ε, και συνέχιση των συζητήσεων έτσι ώστε ε, τα, στα μέσα 2020 να μπορέσουμε να ψηφίσουμε ε, ομοφόνος, διότι χρειάζεται ομοφωνία, το τελικό κείμενο. Ε, το άλλο που θα ήθελα να αναφέρω είναι οι εργασίες για τη δημιουργία στόχων για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030. Ε, θέλουμε να ενισχύσουμε το πολιτικό πλαίσιο για την πολιτική χρήση της ενέργειας, της ανανεώσιμης πηγές ενέργειας, τις εκπομπές αερίων ε, πέρα από το 2020 με νέους στόχους για το 2030. Κατά κάποιο τρόπο αυτό έχετε να επαναλάβει, να αντιγράψει το σύστημα που ε, έχουμε θεσπίσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου έχουμε στόχου για το 2030. Στα πλαίσια λοιπόν τη ίδια λογική, πέρυσι το 2018 ενέκρινε μια σύσταση η ενεργή κοινότητα για την προπαρασκευή για την ανάπτυξη σχεδίων ενέργειας για το κλίμα. Θα τα γνωρίζετε αυτά, διότι αυτό ακριβώς κάνουμε και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου επίσης ξεκινήσαμε ε, πριν τον κανονισμό για τη διακυβέρνηση της ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, είχαμε κατευθυντήρες γραμμές ε, για, μια, για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα εντός της ενεργής κοινότητας θα πρέπει να καλύπτουν την περίοδο από το 2021 έως το 2030 και να ανοίγει ένα δρόμο, ανοίγουν ένα δρόμο για να επιλεχθούν οι στόχοι που έχουν ε, συμφωνηθεί για το 2030 με βάση αυτό που θα πρέπει να φέρει ως αποτέλεσμα το καθένα από συμβαλόμενα μέρη, την baseline δηλαδή, και βεβαίως πρέπει να υπάρχει μια προοπτική, προοπτική και με ορίζοντα το 2050 για να υπάρχει μια συνέπεια με τους μακροπρόθεσμους στόχους, τους πολιτικούς στόχους που έχουμε θέσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών και σε επίπεδο ενεργειακή κοινότητα. Ε, τα σχέδια σχεδίων, τα σχέδια προγραμμάτων πρέπει να υποβληθούν έως ε, το Μάρτιο του 2020 στη Γραμματεία και στη συνέχεια η Γραμματεία θα εκδώσει κάποιες γνωμοδοτήσεις για αυτά τα ενεργειακά σχέδια όπως έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή και με τα προσχέδια ε, των κρατών μελών νωρίτερα φέτος. Τα τελικά σχέδια θα υποβληθούν στα τέλη του 2020 λαμβάνοντας υπόψη ε, βεβαίως τα σχόλια της γραμματείας πέρσι τον Νοέμβριο η Υπουργική Σύνοδος ενέκρινε κάποιες γενικές κατευθυντικές γραμμέ πολιτική για του στόχου του 2030. Σύμφωνα με αυτέ τις κατευθυντικές γραμμές, οι στόχοι του 2030 θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με του στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση του 2030, δηλαδή θα πρέπει να είναι εξίσου φιλόδοξα για συμβαλόμενα μέρη και θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη βεβαίω οι κοινωνικο-οικονομικέ διαφορέ, οι τεχνολογικέ εξελίξει, ε, και τη Συμφωνία των Παρισίων για τη κλιματική αλλαγή. Ε, πρέπει να υπάρχουν στόχοι για όλα τα συμβαλώμενα μέρη, ε, στο σύνολό τους, αλλά και ατομικά. Και εκεί ενδεχομένω να έχουμε και διαφορετική προσέγγιση, διότι όπω γνωρίζετε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ό,τι φορά την αποδοτική χρήση τη ενέργεια και τα ανανεώσιμα, συμφωνήσαμε μόνο για ευρωπαϊκού στόχου και όχι για εθνικού θεσμευτικού στόχου. Το Υπουργικό Συμβούλιο εξέφρασε επίση την πρόθεσή του να συμπεριλάβει στόχους του 2030 όταν θα συμφωνηθούν ε, στο νομικό πλαίσιο της ενεργειακής κοινότητας με τροποποίηση της οδηγίας για την αποτυχία της ενέργειας, ε, για τι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για τη νέα διακυβέρνηση όταν αυτά θα εφαρμοστούν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσφατα ολοκληρώσαμε την προσέγγιση μας από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής εν ώψη των στόχων του 2030 στην ενεργειακή κοινότητα, ο στόχο μας είναι επί τη βάση των αποτελεσμάτων ενό μια νέας έρευνας να προτείνουμε στόχους αρχές 2021. Ε, ο στόχος είναι να ξεκινήσει η μελέτη τον Απρίλιο του 2020. Εν τω μεταξύ, και για να μην χάνεται έτσι ε, το momentum. Η πρόταση στην Υπουργική Συνόδο είναι να εγκρίνουμε ένα οδικό χάρτη όπου θα δεσμεύεται η ενεργειακή κοινότητα ε, για πιο μακροπρόθεσμους στόχους, τον στόχο της κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050, εφόσον βέβαια μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για τέτοιου μακροπρόθεσμους στόχους ε, έω το τέλος του έτου στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτά ε, εν συντομία ε, αυτά τα οποία ήθελα να αναφερθώ, τα βασικά δηλαδή ζητήματα στη σχέση μας με την ενεργή κοινότητα και βεβαίω είμαι στη διαθεσία για να απαντήσω οποιοδήποτε ερώτημα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you so much, Ms. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πένιο για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εισαγωγή που κάνατε. Και τώρα θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Έχουμε τον κύριο Μπούζεκ ως εισηγητή, την κυρία Καρβάλιο από το ΕΛΚ. Δεν ξέρω ποιος θέλει πρώτος να μιλήσει ε, εξ του ΕΛΚ. Παρακαλώ, η κυρία Καρβάλιο. Ευχαριστώ, κυρία Παολαπίνιο. Ε, χαίρομαι που σας βλέπω. Είμαστε φίλες. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε πώς γίνεται αυτός ο εξυγχρονισμός της ενεργειακής κοινότητας και ότι εισάγεται διάφορες συμφωνίες και φιλοδοξίες και στόχους και για τις χώρες γειτονίας. Επίσης, η ενίσχυση της εφαρμογή της υλοποίησης είναι πολύ σημαντική και η αμοιβαιότητα είναι κάτι το πολύ σημαντικό που εισάγεται εδώ. Συμφωνώ απόλυτα με τους στόχους. Και θέλω να σας θέσω δύο ερωτήσεις. Πρώτη, είναι πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια για αυτές τις χώρες όσον αφορά την οικοδόμηση δυνατοτήτων, αλλά από πρακτικής άποψης ποιο ήταν το αποτέλεσμα και η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην ενεργειακή πολιτική και στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση είναι ότι στις διαπραγματεύσεις για το κλίμα είναι κομμάτι ενός ε, διαφορετικού συνόλου. Ε, βλέπουμε πως υπάρχει δυνατότητα σε αυτήν την αναθεώρηση να υπάρξει μια καλύτερη σύνδεση στις διαπραγματεύσεις για το κλίμα ε, με τις χώρες αυτές. Κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ θετικό για την Ένωση, γιατί έτσι θα είχαμε περισσότερη συγκέντρωση κρίσιμης μάζας, ακόμα και αν είναι άτυπη συνεργασία. Και αυτό γιατί υπάρχει πάντοτε διαβούλευση για τα κράτη-μέλη της Ένωσης, ώστε να μιλάμε με μια φωνή. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να έχουμε μια συμφωνία και με αυτές τις χώρες, γιατί έχουμε τις ίδιες φιλοδοξίες και στόχους, εάν συμφωνήσουμε. Θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε μια δεύτερη κοινή φωνή στις διαπραγματεύσεις για το κλίμα. Και αυτό θα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Καρβάλιο. Κάποιος από τους σοσιαλιστές θέλει να πάρει το λόγο. Η Ρινιού, παρακαλώ. Ο κύριος Φλέγκο. Σας ευχαριστώ για αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα που θέσατε σήμερα στην ημερήσια διάταξη. Γνωρίζουμε όλοι πόσο μεγάλη είναι η σημασία αυτής τη κοινότητας ενέργειας. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση σε προσιτή ενέργεια με βάση τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Αυτό όμω που είναι εξίσου σημαντικό είναι πως η ενέργεια είναι σημαντική ναι μεν για την βιομηχανία αλλά και για τον ευρύτερο πληθυσμό. Η ενέργεια είναι σημαντική για τη βιομηχανία βιομηχανία, ναι, και ε, σε αυτό το πλαίσιο αναφέρομαι στον ανταγωνισμό. Στον ανταγωνισμό της ε, βιομηχανίας, ε, γιατί η τιμή της ενέργειας είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την πράσινη ενέργεια, να θυμίσω τη Συμφωνία του Παρισιού και την ανάγκη να συμμορφωθούμε προς τους στόχους αυτής της συμφωνίας. Ναι, αλλά ωστόσο πιστεύω πως οι στόχοι των κρατών μελών θα πρέπει να ακολουθήσουν με τη σειρά τους. Δεν αρκεί δηλαδή να φτιάχνουμε σχέδια, πρέπει και να τα υλοποιήσουμε στη συνέχεια. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο προϋπολογισμός ε, 2021 με 2027 θα πρέπει επίσης να ακολουθήσει αυτή την ενεργειακή μετάβαση με τα κατάλληλα κονδύλια. Διερωτώ με λοιπόν εάν έχει, είστε της ίδιας άποψης. Γιατί τα χρήματα είναι σημαντικά, οι νομοθεσίες είναι σημαντικές και όλοι μαζί αποτελούν τους σημαντικούς ε, παράγοντες ε, για μια επιτυχή μετάβαση προς πράσινη ενέργεια, χωρίς ωστόσο να να χάσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. κύριος Νίνιστο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, είναι μια ευκαιρία για να συζητήσουμε για θέματα που είναι προβληματικά στη συνεργασία και αυτό έχει να κάνει με τις συμβάσεις και με την ε, υλοποίηση των ε, υφιστάμενων δεσμεύσεων καθώς και με τους στόχους όσον αφορά την ε, αναχέτηση των κλιματικών αλλαγών. Η ομάδα μας λοιπόν έχει αμφιβολίες. Ε, δεν υπάρχει μηχανισμός ε, επιβολής σε περίπτωση μη εφαρμογής. Υπάρχει επίσης έλλειψη διαφάνειας και ακόμα και διαφθορά εκτεταμένη σε κάποιες από τις συνυπογράφουσες χώρες. Δεν γίνεται λόγο ΣΟΕΔΕ για την ε, συμμετοχή των ΜΚΟ σε αυτήν την προσπάθεια. Ποιες προβλέψεις λοιπόν ε, ε, έχετε κάνει για την εφαρμογή όλων αυτών εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου. Έχετε συμφωνήσει για κάποιο σύστημα ελέγχου που να είναι αποτελεσματικό ώστε να εξασφαλίσουμε την επίτευξη των στόχων και την τήρηση των δεσμεύσεων. Τώρα, Υπάρχουν πάντοτε παραβάσεις, ας πούμε, ε, ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες που δεν ε, σέβονται τις σχετικές νομοθεσίες, ε, δεν εφαρμόζονται ούτε οι στόχοι για την ενεργειακή επάρκεια. Επίσης, εφαρμόζεται η δυνατότητα για περιβαλλοντικές, ε, ε, περιβαλλοντικά έργα. Ας πούμε, ένας νέος ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή στη Βοσνία. Πώς σκοπεύετε λοιπόν να ενεργήσετε για την τήρηση αυτών των προγραμμάτων ενέργειας, των σχεδίων ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ. Από την ομάδα ID, ο κύριος Πόρχε. Σας ευχαριστώ. Τα κράτη-μέλη προσπαθούν να επιτύχουν τις μηδενικές ε, εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα, ενώ εφόσον μάλλον ε, ε, κάνουμε τέτοιου είδους συμβάσεις με τρίτες χώρες αναμένεται να ακολουθήσουν το ίδιο μονοπάτι. Ωστόσο, ο τομέας αυτός ε, στο Κωσυφοπαίδιο, στη Βοσνία Ριζεγοβίνη και στη Βόρεια Μακεδονία δεν φαίνεται να πληρούνται αυτές οι προδιαγραφές. Τα Δυτικά Βαλκάνια επίσης στηρίζονται από κινέζικες επενδύσεις. Θα ήθελα να ακούσω κάποιο σχόλιο από την Κομισιόν για αυτό το ζήτημα. Στην παρέμβασή σας αναφέρατε ότι ο γενικός στόχος είναι η ανάπτυξη του ανταγωνισμού. Θα ήθελα να γνωρίζω αν έχετε ενδείξεις ε, ε, σχετικά Ε, σχετικά με την επίδραση αυτής της συμφωνίας ε, ε, στους γενικούς πληθυσμούς. Ευχαριστώ. Αν θέλετε να απαντήσετε στην πρώτη, στον πρώτο αυτό γύρο ερωτήσεων και μετά θα ακούσουμε και άλλες ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ όλους. Κυρία Καρβάλιο, όντως, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι μέσω της ενεργειακής κοινότητας θα συμβάλλουμε επίσης στην κοινή φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ε, συνεταίρους της. Στη, τα συμβαλόμενα μέρη στην ε, Συμφωνία του Παρισιού και στην εφαρμογή της ε, έχουν εκεί δεσμευθεί και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με τους εταίρους μας της, κοινότητας, ε, της ενεργειακής κοινότητας είναι να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε νομοθεσία που να περιλαμβάνει και την κλιματική νομοθεσία από πλευρά της Ένωσης και με αυτό σαφώς θα έχουμε τους εταίρους μας με την πλευρά μας, όχι μόνο με τη ρυθμιστική πλευρά, αλλά εφαρμόζοντας τους ίδιους κανόνες αναμένουμε ότι η συνέπεια θα είναι και η πολιτική έγκριση και στήριξη της προσπάθειας αυτής με την έννοια ότι θα προχωρούν όλα προς την ίδια κατεύθυνση όσον αφορά τη Συμφωνία του Παρισιού. Πιστεύουμε λοιπόν πως έτσι θα μπορέσουμε έμεσα να βοηθήσουμε ώστε να έχουμε εταίρους που θα, μιλάμε, θα μιλάνε ακριβώς με μια φωνή όσον αφορά ε, την ε, ε, ενέργεια. Τώρα, έχουμε δει πρόοδο. Ας πούμε, τώρα συζητάμε τους στόχους 2030 για την ενέργεια και το κλίμα με την συμβαλόμενα μέρη της ενεργειακής κοινότητας, αλλά ωστόσο πρέπει να τονίσουμε πως ήδη εφαρμόζεται το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο για το 2030, όπου όντως υπάρχει πρόοδος σε διαφορετικά επίπεδα και με διαφορετικό ρυθμό. Αλλά σίγουρα υπάρχει θετικός αντίκτυπος ε, από το γεγονός ότι αυτά τα συμβαλώμενα μέρη έχουν υιοθετήσει το ευρωπαϊκό και εκτιμένο επίσης μέσα στην ενεργειακή κοινότητα με τους ίδιους κανόνες, τις ίδιες διατάξεις και παρά το γεγονός ότι ε, ε, όσον αφορά την επιβολή εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια κενά. Μπορούμε να δούμε λοιπόν ποιος είναι ο θετικός αντίκτυπος των κανόνων αυτών. Τώρα, όσον αφορά τον αντίκτυπο της ενεργειακής κοινότητας στην ε, βιομηχανία στον κόσμο και τη σημασία του να έχουμε στόχους αλλά επίσης να τους εφαρμόζουμε. Εμείς επιδιώκουμε μια παρόμοια προσέγγιση όπως αυτή που ακολουθήσαμε στο, στην Ένωση για το 2030. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο πρόκειται για μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω που λαμβάνει υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες των συμβαλόμενων μερών και αυτό θα οδηγήσει στη δημιουργία είτε ενός συλλογικού στόχου για ολόκληρη την ενεργειακή κοινότητα, είτε σε μονομένους ατομικούς μάλλον στόχους. Όπως ε, είπα και προηγουμένως, η ιδέα είναι να μπορέσουμε σε αυτή τη βάση να αντικατοπτρίσουμε τις εθνικές ιδιαιτερότητες. μέσα σε αυτή την ομάδα των συμβαλωμένων μερών. Σε κάθε περίπτωση αυτό που ήδη βλέπουμε και από τις συζητήσεις είναι ότι υπάρχει η προσχώρηση στην αρχή της εθνικής ταυτότητας και των εθνικών σχεδίων όπου θα ζητήσουμε τους στόχους αλλά και πολιτικές και μέτρα για το πώς σκοπεύουν να ε, υλοποιήσουν αυτούς τους στόχους. Να μην έχουμε δηλαδή μόνο θεωρίες και φιλοδοξίες αλλά να έχουμε και να γνωρίζουμε πώς τα συμβαλόμερα να μέρη σκοπεύουν να υλοποιήσουν στην πράξη αυτούς τους στόχους. Ο μηχανισμός επιβολής είναι ένας από τους τομείς που όντως χρειάζεται βελτίωση και γι' αυτό και είναι και ένας από τους τομείς που τώρα ε, μας απασχολεί στη μεταρρύθμιση της κοινότητας ενέργειας ώστε να μετρήσουμε τις ε, επιπτώσεις ε, της διαδικασίας ε, υπό τη συνθήκη, να ενισχύσουμε το ρόλο των ανεξάρτητων νομικών χρηματοδοτήσεων της Συμβουλευτικής Επιτροπής, να εισάγουμε πρόστιμα σε περίπτωση που δεν συμμορφούνται προς το κεκτημένο της ενεργειακής κοινότητας, ένα τρόπος όπου προσπαθούμε όντως να ενισχύσουμε αυτό το τομέα που βλέπουμε πως υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Τώρα, για τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, ε, όντως δεν εφαρμόζονται απαραίτητος οι ευρωπαϊκοί κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, που σημαίνει ότι και πάλι οι κρατικές ενισχύσεις είναι μια από τις πτυχές που εξετάζονται στο πλαίσιο αυτής της μεταρρύθμισης. Η ιδέα είναι να ενισχυθεί η εφαρμογή των κανονισμών για τις κρατικές ενισχύσεις ε, αναφερόμενοι συγκεκριμένα στο κεκτημένο, να προσπαθήσουμε δηλαδή να ωφεληθούμε από το μέγα δυναμικό που εξακολουθεί να υπάρχει στα συμβαλόμενα μέρη της ενεργειακής κοινότητας. Και τέλος, και κατά κάποιο τρόπο νομίζω ήδη το αναφέρα αυτό, ότι αναγνωρίζουμε δηλαδή τις εθνικές ιδιαιτερότητες των συμβαλόμενων μερών, το γεγονός ότι πολλοί εξ αυτών όντως εξαρτώνται από τον άνθρακα ως βασική, ε, βασικό πόρο, βασικό κομμάτι του ενεργειακού μείγματος ε, και αυτό είναι κομμάτι της διαδικασίας, η σταδιακή πάυση της χρήσης άνθρακα προβλέπεται για όλα τα συμβαλόμενα μέρη. Ευχαριστώ πολύ για αυτό τον ε, πρώτο γύρο και τώρα μπορούμε να επιστρέψουμε και να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μπουζά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ επίσης που μας παρουσιάσατε τα θέματα αυτά και θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ενεργειακή κοινότητα παραμένει ένα πολύ σημαντικό θέμα όχι μονάχα για τα συμβαλόμενα μέρα αλλά και για τα κράτη-μέλη και έτσι ε, λοιπόν μπορούμε να πιάσουμε δύο τριγώνια με ένα σβαρό δύο τριγώνια. Ε, μπορούμε να φέρουμε γειτονικέ χώρε πιο κοντά στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν ε, να πω ε, έχουμε την έκθεση Μια Ενεργειακή Ένωση για το μέλλον. Συγχαρητήρια λοιπόν για το ότι εφαρμόσατε βήμα-βήμα όλα τα θέματα τα οποία αναφέρθηκαν στη συγκεκριμένη έκθεση. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως να μην είναι πάρα πολύ γρήγορη, αλλά είναι πάρα πολύ ακριβής και ύστερα από κάποια χρόνια μπορούμε να εφαρμόσουμε ό,τι έχουμε προβλέψει για ένα τέτοιο θέμα. Και επίσης ε, θα ήθελα να κάνω άλλο ένα σχόλιο για τα τελευταία τρία χρόνια. Ε, συνδιοργανώνω ε, την ε, Επιτροπή Συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την, με την, Ευρωπαϊκή κοινότητα, την Ενεργειακή Κοινότητα τον Απρίλιο θα έχουμε την επόμενη συνάντησή μας. Η Ολομέλεια είναι στις 12 Δεκεμβρίου, όπως είπατε και εσείς. Και θα ήθελα να πω στους συναδέλφους, σας καλώ να παραβρεθείτε σε αυτές τις συναντήσεις. διότι θα έρχουν ε, εκπρόσωποι των κοινοβουλίων από τα συμβαλόμενα ε, μέρη 10-12 αντιπρόσωποι ε, θα είναι και μερικές φορές και από άλλες πλευρές, από τη δική μας πλευρά έχουμε μονάχα έναν-δύο αντιπροσώπους και αυτό είναι άδικο, οπότε θα ήθελα να σας παρακαλέσω να έρθετε και να το συζητήσουμε με τους συναδέλφους από τα συμβαλόμενα μέρη. Δύο ερωτήσει τώρα. Ε, αρχικά, πώ η Επιτροπή θα διασφαλίσει ότι οι ε, διαπραγματεύσει ε, για τι ε, ε αλλαγέ των συνθήκων δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα σε χώρε όπω είναι η Σερβία και το Κόσοβο, όπου υπάρχουν προβλήματα και πώ ε, και ε, τι συμβαίνει ε, σε περίπτωση που δεν θέλουν όλα τα συμβαλόμενα μέρη να υπογράψουν τη νέα συνθήκη. Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο. Αναφέρατε επίσης την ενίσχυση των κανόνων όσον αφορά την ενημέρωση για τις κρατικές ενισχύσεις, κάτι το οποίο το συζητήσαμε σε επίπεδο ε, σε υψηλό επίπεδο, αλλά επίσης ε, και η κοινωνία των πολιτών ε, ζητά να συμμετάσχει στην, στην όλη διαδικασία. Έτσι λοιπόν πώς θα διασφαλίσετε την εφαρμογή των κανόνων για, την, για τις κρατικές, για τις Έχουμε για παράδειγμα ε, τις ε, κινέζικες επενδύσεις ε, σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από άνθρακα στην Βοσνία, το οποίο μπορεί να αποτελέσει ένα πρόβλημα για εμάς και για, τόσο για το Κοινοβούλιο όσο και για τα υπόλοιπα συμβαλόμενα μέρη. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι που μας ε, παρουσιάσατε καθώς επίσης και για όλες σας τις δραστηριότητες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπούσεκ. Ακολουθεί ο κύριος Κέλλη από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά το, τους ε, στόχους την προηγούμενη εντολή του Κοινοβουλίου, την, ε, την προηγούμενη περίοδο, ε, ασχοληθήκαμε με θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενεργειακή αποτελεσματικότητα κτλ. Ε, τώρα λοιπόν, αν θέλουμε να αυξήσουμε την φιλοδοξία, είναι κάτι το οποίο αγαπούν οι πολίτες, την αύξηση των φιλοδοξιών, πολύ συχνά οι στόχοι αυτοί τίθενται από ανθρώπους που βάζουν σε άλλους να τους εφαρμόσουν τι θα γίνει λοιπόν με τα κράτη-μέλη τα οποία τώρα ολοκληρώνουν ε, τα εθνικά τους ε, σχέδια για την ενέργεια και το, ε, κλίπα, για το κλίμα. τι θα γίνει, θα περιμένουμε, διότι όλα αυτά βασίζονται σε στόχους τους οποίους θέσαμε τα τελευταία χρόνια. Και δεύτερον, και συμφωνώ απολύτως με όλους όσους είπαν ότι οι στόχοι έχουν ε, συμφωνηθεί. Αυτό είναι ένα θέμα, αλλά η εφαρμογή του είναι κάτι εντελώ ε, διαφορετικό. Δεν έχουμε εθνικά δεσμευτικού ε, στόχου αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να έχουμε δεσμευτικούς στόχους και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. και τα σχέδια αυτά θα παρακολουθούνται σε ετήσια, σε διετή ε, βάση ή ε, μετά από 4-5 χρόνια θα δούμε κάποιες ε, χώρες που έχουν ξεφύγει από τους στόχους, θα βρίσκουν διάφορες δικαιολογίες που δεν εφαρμόσαν τους στόχους, διότι αν οι κυβερνήσει δεν έχουν ένα κίνητρο ώστε να λάβουν μέτρα και να έχουν και την απαραίτητη υποστήριξη, τότε δεν πρόκειται να ε, πραγματοποιήσουν τους ε, στόχους αυτούς ε, και φοβάμαι ότι πολλοί από αυτούς τους στόχους θα είναι απλά μια επιθυμία και τελικά και εν τέλει δεν θα συμβεί τίποτα. Σε αιτήσια βάση τώρα θα ήθελα να δω πώς θα κάνουμε την πρόοδο που χρειάζεται να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κέλλη. Η κυρία Πάουλους ε, από τους ε, Πράσινους, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να επαναλάβω ένα ε, ρόλο είπατε ότι θα ενισχυθεί ο ρόλος των ενδιαφερόμενων μερών ε, του ε, Συμβουλευτικού Συμβουλίου, όμως εγώ θα ήθελα να, πείτε κάποιες, να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με το τι εννοείται όταν λέτε θα ενισχυθεί ο ρόλος τους, διότι δεν είναι ένα μετρήσιμο στοιχείο. Ε, και δεν ε, δίνει πληροφορίες σχετικά με την όλη διαδικασία. Και το δεύτερο τώρα ερώτημα είναι Ε, δεν κατάλαβα ακριβώς ε, τι θα γίνει με τις διαδικασίες επιπαραβάση. Ε, έχει όλο αυτό να κάνει με την απόφαση ε, του Συμβουλίου σχετικά με τις ε, προοπτικές διεύρυνσης που δημοσιοποιήθηκε προσφάτως. Ίσως λοιπόν οι απαιτήσει να μην είναι τόσο ισχυρές όσο θα έπρεπε να ήταν. Ευχαριστώ κύριε Παύλος. Και τέλος ο κύριος Κουμπίλιους. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ως ε, νέος ε, ευρωβουλευτής θα θέσω ένα ερώτημα που ίσως να φανεί αφελές. Ναι, η ενεργειακή ε, κοινότητα ε, έχει αρκετά ε, θετικά. Όμως ένα παράδειγμα τώρα, η Ουκρανία. Το ερώτημά μου είναι πώς θα περιγράφατε τι όφελος φέρει η ενεργειακή κοινότητα για την Ουκρανία, η οποία θα πρέπει να αναθεωρήσει τον ενεργειακό της τομέα, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν ε, και αρκετά σοβαρά ζητήματα όπως είναι η ε, ασφάλεια του εφοδιασμού ή διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία σχετικά ε, με την μεταφορά. Βλέπουμε διάφορα θέματα να συζητούνται. Βλέπουμε τι επηρεάζει την Ουκρανία για να μπορέσει να αναθεωρήσει τον ενεργειακό της τομέα. Και παράδειγμα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ε, απαιτεί ε, μεγάλες μεταρρυθμίσεις όσον αφορά την τιμολόγηση του ενεργειακού τομέα, αλλά όχι εξαιτίας της ενεργειακής κοινότητας. Έχουμε για παράδειγμα την ε, Gazprom η οποία δεν περνάει μέσω της ενεργειακής κοινότητας. Το απλό μου ερώτημα λοιπόν είναι το πώς θα περιγράψουμε τα κίνητρα ε, για την ενεργειακή κοινότητα, ούτως ώστε χώρες όπως είναι η Ουκρανία να ε, προχωρήσουν και να έχουν κάποιο πραγματικό όφελος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίλιους. Κύριε Πινιούς, έχετε τον λόγο να απαντήσετε σε αυτές τις ε, ερωτήσεις και να ολοκληρώσετε. Κύριε Μπούζακ, έχετε απόλυτο δίκιο. Και με βάση τις ε, τεχνικές συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις ε, θα χρειαστούμε και ε, πολιτικό κεφάλαιο και διπλωματία, διότι φυσικά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το γεγονός ότι μπορεί να υπάρξουν διαφορετικά εθνικά συμφέροντα μεταξύ των συμβαλόμενων μερών κάτι ε, το οποίο θα ε, δημιουργήσει προκλήσεις ε, στην ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης και φυσικά εργαζόμαστε πάνω σε αυτά τα θέματα μέσω της ε, διπλωματικής οδού για να μπορέσουμε να αποφύγουμε ε, τυχόν τέτοιες ε, διαμάχες οι οποίες να κρατήσουν όμοιρο την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης. Είχαμε μια συνάντηση υψηλού επίπεδου όπου ο στόχος είναι να διασφαλίσουμε την επίτευξη συμφωνίας τον Δεκέμβριο εξετάζουμε όλες τις εναλλακτικέ ε, θέσεις, ε, τους ε, συμβιβασμούς για να μπορέσουμε ότι εν να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι εν τέλει θα υπάρξει συμφωνία. Τώρα όσον αφορά την εφαρμογή, μπορούμε να εξετάσουμε την εφαρμογή μονάχα από ρυθμιστικής πλευράς, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως και θα πρέπει να γίνουν περισσότερα πάνω σε αυτό. Το απλό ε, θέμα είναι ότι υπάρχει αυτή η ε, κοινότητα η οποία προσφέρει την ε, δυνατότητα και για πολιτικές συζητήσεις με αποτέλεσμα να υπάρχει μια θετική πίεση και εντός των ε, συμβαλόμενων μερών της ενεργειακής κοινότητας αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά υπάρχει η όρεξη να ακολουθούν οι κανόνες και αυτό ε, φυσικά απαντά και το τελικό ερώτημα Αν έχουμε ένα σταθερό νομοθετικό πλαίσιο, αυτό αποτελεί το κλειδί για την προσέλκυση επενδύσεων και ταυτόχρονα ε, βοηθά στο να παραδώσουμε ε, και άλλους ε, στόχους. Και παράδειγμα, όταν μιλάμε λοιπόν για την Ουκρανία, προφανώς αυτό είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η Ουκρανία αντιλαμβάνεται την ανάγκη να συμμορφωθεί. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν το δούνου του και όχι η ενεργειακή κοινότητα, αλλά πιστεύω πιστεύω ότι εν τέλει ήταν συνδυασμό παραγόντων και δεν μπορούμε μονάχα μέσω του ε, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να ε, προωθήσουμε αυτές τις ε, μεταρρυθμίσεις. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σταθερό περιβάλλον το οποίο θα ε, προσελκύσει επενδυτές, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τις υποδομές για το φυσικό ε, αέριο είναι λοιπόν ένας ε, συνδυασμός παραγόντων και αυτό είναι και το μεγάλο όφελος της ε, διεθνούς ε, συνεργασίας και μέσω της δικής μας συνεργασίας με άλλους θεσμούς και έτσι λοιπόν μπορούμε να διασφαλίσουμε μια συνθήκη που κερδίζουν όλοι. Τώρα για τον κύριο Κέλλη. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα ερώτημα το οποίο αφορά περισσότερο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και όχι την ενεργειακή κοινότητα. Τι γίνεται αν αυξήσουμε τις ε, φιλοδοξίες. Φυσικά και τα σχέδια ε, για το κλίμα και την ενέργεια θα κοινοποιηθούν αρχές της επόμενης την επόμενη χρονιά ε, στην Επιτροπή και ε, θα ε, συγκριθούν με τους στόχους για το 2030. Οι στόχοι του 2030 της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ελάχιστοι στόχοι. Μιλάμε για 32% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό όμως δεν αποτρέπει τίποτα τα κράτη-μέλη ε, το να έχουν πιο φιλόδοξους ε, στόχους ε, και είχαμε κράτη-μέλη που στα προσχέδιά τους έχουν ήδη προσχεθεί περισσότερα από αυτά τα οποία απαιτούνται για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων. Σε κάθε περίπτωση, είτε αυξηθεί η φιλοδεξία είτε όχι, οι στόχοι του 2030 αποτελούν ε, το σημείο για την παράδοση οποιονδήποτε άλλων στόχων. Θα ε, αξιολογήσουμε τα σχέδια αυτά σε σχέση με τους στόχους του 2030. Τώρα, όσον αφορά την παρακολούθηση, θα δούμε, θα παρακολουθούμε ανά δύο χρόνια το πώς εφαρμόζονται οι στόχοι αυτοί επισήμως μέσω μιας έκθεσης η οποία θα κοινοποιείται και σε εσάς και ε, τότε θα εξετάζουμε το πού βρίσκονται τα κράτη-μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των ε, στόχων τους ε, και τις συνεισφορές που έχουν παρουσιάσει στους στόχους για την ενέργεια και το κλίμα. Τώρα όσον αφορά το ζήτημα της εφαρμογής και ότι θα πρέπει να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι πάνω σε αυτό. Είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται ακόμα, διότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσει. Έτσι λοιπόν δεν μπορώ να ξέρω ποια θα είναι το τελικό αποτέλεσμα των ε, διαπραγματεύσεων. Όμω ε, θα υπάρχουν ε, σίγουρα μηχανισμοί οι οποίοι ε, δεν θα είναι τόσο εθελοντική διάσταση, θα, έχουν, ε, θα είναι δεσμευτικοί. Ε, ελπίζω να υπάρξει ένα ξεκάθαρο κείμενο για να μπορέσουμε ξεκάθαρα να πούμε τι θα συμπεριλαμβάνεται πάνω σε αυτό. Και όσον αφορά την ερώτηση του κυρίου Κουμπίλιους, πιστεύω ότι ήδη απάντησα, απαντώντας και την ερώτηση του κυρίου Μπουζέκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πίνιος για αυτήν την ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή Ήτρε για αυτό το σημαντικό θέμα που αφορά την ενεργειακή κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε σήμερα και μας παρουσιάσατε τη θέση σας. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα ήθελα να καλέσω τον ε, κύριο Τζέρμι ε, Τζόφρι, ε, τον κύριο Τζαν Σόμπλουμ και τον κύριο Ιγνέση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο σημείο 6, 5 της σημερισίας διάταξης, ανταλλαγή απόψεων με τον επικεφαλής της, του οργανισμού BEREC 2019, καθώς επίσης και τον επερχόμενο πρόεδρο του 2020 ε, κύριο ε, Σιόμπλομ, καθώς επίσης και τον Διευθυντή της Υπηρεσίας για την Υποστήριξη του Μπέρεκ, κύριο Ιγνέση. Παρακαλώ. So, was a leak. Ο λοιπόν, Νίτρε είναι η ομάδα η οποία είναι υπεύθυνη για τι τελευταίε εργασίε σχετικά με τον κώδικα του προκάτου επικοινωνιών που θα πρέπει να μεταφερθεί έω τον Δεκέμβριο του 2021 ε, καθώς και την αναθεωρημένη ε, τον κανονισμό Μπέρεκ που τέθηκε σε ισχύ πέρυσι. Και βεβαίω αναμένουμε να ακούσουμε από τον πρόεδρο, τον κύριο Γκάτφρι, πώ λειτουργεί το Μπέρεκ σε ό,τι αφορά τι εργασίε για τον κώδικα τηλεπικοινωνιών ε, ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών και ο κύριος Σύπλων που θα είναι πρόεδρος για το 2020 να μας πει πώς αναμένει να προχωρήσει η όλη διαδικασία. Ε, να ακούσουμε τον κύριο Γκόρτσερ και τον κύριο Εγνάση επίσης για τις πρώτες εμπειρίες τους με τον νέο κανονισμό Derek λαμβάνοντας υπόψη όλες τις εργασίες που έχουν λάβει χώρα σε αυτή την Επιτροπή. Το Μπέρεκ παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο ε, για την περιαγωγή, για την κυβερνοασφάλεια, ε, πολύ σημαντικά ζητήματα ε, για τα οποία θα θέλαμε επίσης να ενημερωθούμε. Έχουμε περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο προβλέψει για αυτό το θέμα στη Μέση Διάταξη, οπότε θα ήθελα να δώσω το λόγο ευθύς αμέσως στον κύριο Godfrey. Ε, καλώς ήρθατε, αναμένουμε την παρουσίασή σας. Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα σε όλους εισαγωγικά να σας πω ότι ε, κάποιος μου παρουσίασε ως πρόεδρο του και το 2019, αλλά είμαι και επίτροπος της Κόμνεκ του Ρυθμικής Αρχής της Ιρλανδίας. Ο Σάνφος είναι ε, επικεφαλή του PTX, του Σουηδίου, της Σουηδική Ρυθμικής Αρχή και του χρόνου θα είναι πρόεδρο του Μπέρεκ. Και ο Λάσλο είναι ο διευθυντής του γραφείου του Μπέρεκ. Ε, Δυστυχώς δεν μπορούμε να δείξουμε τις διαφάνειες. Ε, θα μιλήσω για τρία σημεία στην παρουσίασή μας. Για τα νέα μέλη πρώτα απ' όλα. Εγώ και ο Λάσλο θα σας παρουσιάσουμε το έργο του Μπέρεκ, το ρόλο του Μπέρεκ και του γραφείου Μπέρεκ. Στη συνέχεια ο Νταν θα μιλήσει για κάποια ενδιαφέροντα ζητήματα, τον κώδικα, τι έχουμε κάνει για τον κώδικα, την περιαγωγή, την κυβερνοασφάλεια. Στη συνέχεια θα μιλήσω για το 5G ε, και το, το ανοιχτό ίντερνετ και τα νέα ζητήματα που προκύπτουν στα πλαίσια των, των ε, προτεραιοτήτων της Νέας Επιτροπής για μια Ευρώπη που θα είναι έτοιμη για την ψηφιακή εποχή. Σε ό,τι αφορά το ρόλο του Μπέρεκ υπάρχουν τρία πράγματα που κάνει τον Μπέρεκ. Πρώτον, είμαστε υπεύθυνοι να εξασφαλίσουμε μια συνεπή εφαρμογή ε, της νομοθεσίας πολιτερονικών επικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό, όπως είπε ο κύριος Πίτερσον, περιλαμβάνει κάποιες λεπτές γραμμές. Υπάρχουν 11 κατευθυντές γραμμές που ε, θα εκπονήσει το ΜΠΕΡΕΚ κατά την εφαρμογή του νέου κώδικα. Έχουμε όμως γραμμές για την περιαγωγή, για την εφαρμογή του κανονισμού για το ανοιχτό ίντερνετ, ε, το ανοιχτό διαδίκτυο, ατύπως ανταλλάσσουμε εμπειρίες ε, και μεταξύ εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Υπάρχουν προγράμματα κατάρτιση για το προσωπικό και επίση ε, εκθέσεις, βέλτιστες πρακτικές, κοινέ θέσεις ε, κτλ. Το δεύτερο που κάνουμε είναι ότι παράγουμε και κάποιες ιδέες για το μέλλον, την οικονομία των δεδομένων, κάναμε, μια σχετική έκθεση, μια, άλλη έκθεση για το 5G και τι θα πρέπει να γίνει από ρυθμιστικής πλευράς για να επιτρέψουμε την ε, καινοτομία μέσα στο οικοσύστημα του 5G ε, και για τα δίκτυα υψηλής, ε, υψηλών δυνατοτήτων και ποιες είναι οι δυναμικές εκεί και αυτό συνδέεται προφανώς με τους στόχους του κώδικα. Τρίτον, Είμαστε και τεχνικοί σύμβουλοι προς τα θεσμικά όργανα. Ε, το Μπέρεκ λοιπόν με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία παράγει γνωμοδοτήσει ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για περιπτώσεις όπου έχουμε εφαρμοστικές πράξεις ε, και κατά την νομοθετική διαδικασία βέβαια για τον κώδικα και τον κανονισμό Μπέρεκ δώσαμε πληροφορίες και γνωμοδοτήσεις προς τους συνομοθέτες. σας πω ε, λίγο πώς δουλεύουμε και τι είναι αυτό που έχει φέρει ε, την επιτυχία του συστήματος. Υπάρχει ένα συμβούλιο ρυθμιστικών αρχών όπου συμμετέχουν οι επικεφαλή των ρυθμιστικών αρχών των κρατών μελών της Ένωσης. Υπάρχουν όμως και συμμετέχοντες που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ε, από τις χώρες ΕΦΤΑ, από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως το μεγαλύτερο μέρος της δουλειά ε, το κάνουν εκατοντάδε εμπειρογνώμονες ε, οι οποίοι προέρχονται από τις εθνικές αρχές. Υπάρχουν 10 ομάδες ε, εμπειρογνωμόνων για την περιαγωγή, την ανάλυση της αγοράς, στατιστικά. Το καλό με αυτόν τον τρόπο εργασίας είναι ότι αυτέ τις γραμμές που προκύπτουν, οι κοινέ θέσει βασίζονται στις εμπειρίες αυτών που τα χρησιμοποιούν και συνδέεται αυτό και με την πραγματικότητα στην αγορά, επιτόπου, στα κράτη-μέλη, καθημερινά. Επίσης, ε, ε, έχουμε ε, στενή επαφή με τους εμπλεκόμενους φορείς, τον κλάδο, το βιομηχανικό της επιχειρήσης, αλλά και τους καταναλωτές, τους χρήστες δηλαδή ή άλλες βιομηχανίες, όπως η αλλε βιομηχανιε οπω η αυτοκινοβιομηχανια ε, για το πώ θα λειτουργήσουν τα, τα οχήματα, τα οποία θα είναι συνδεδεμένα με το διαδίκτυο. Ε, και ένα άλλο τομέα που αναπτύσσεται είναι η σχέση μα με άλλα όργανα. Πάντα είχαμε στενά όργανα με την πολιτική, με την ομάδα για το ραδιο, ραδιοφωνικό φάσμα. Ε, τώρα πλέον υπάρχουν τα αισθήματα τη ε, κυβερνοασφάλειας, οπότε η ΕΝΙΣΑ είναι ένα ε, εταίρο κλειδί για μας. Έχουμε διασυνδέσεις και με ρυθμιστικές αρχές, με ρυθμιστικά δίκτυα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ανταλλάσσουμε βέλτιστες πρακτικές. Ε, κατά κάποιο τρόπο προωθούμε παγκοσμίω το ευρωπαϊκό μοντέλο τηλεπικοινωνιών ε, και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον ανά τον κόσμο για τις πρακτικές που ακολουθούνται στην Ευρώπη. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον Λάζλο, ο οποίος θα σας μιλήσει για το γραφείο Μπέρεκ. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ήτρε, είναι χαρά μου να σας παρουσιάσω τα βασικά καθήκοντα, της αρμοδιότητες του γραφείου Μπέρεκ και να αναφερθώ ε, στην δομή μας που είναι, δεν είναι μοναδική αλλά δεν είναι και τόσο συνηθισμένη. Το γραφείο Μπέρεκ δημιουργήθηκε ως μια υπηρεσία της Ένωσης για να υποστηρίξει τον Μπέρεκ. Όπως βλέπετε εδώ στον χάρτη υπάρχουν πολλές αποκεντρωμένες ε, ευρωπαϊκές υπηρεσίες σε διάφορους τομείς πολιτικής και το γραφείο Μπέρεκ βρίσκεται στη Ρήγα, στην Λετωνία. Αυτό αποφασίστηκε μετά την έγκριση ε, του προηγούμενου ρυθμιστικού πλαισίου και του κανονισμού Μπέρεκ το 2009. Εδώ και 10 χρόνια λοιπόν περίπου ε, βρισκόμαστε στη Ρήγα και δίνουμε την απαραίτητη υποστήριξη για το έργο του Μπέρεκ όπως μας είπε και ο κύριος Μπέρεκ πριν από λίγο. Στο επόμενο, στην επόμενη διαφάνεια τώρα θα ήθελα να συνοψίσω κάπως ε, τα βασικά καθήκοντα αυτής της μικρής ε, ευρωπαϊκής υπηρεσίας για να καταλάβετε κάπως καλύτερα πώς διευκολύνουμε ως ευρωπαϊκό όργανο το έργο των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το αρχι... Η αρχική ιδέα δημιουργίας της ε, υπηρεσίας υποστήριξης του Μπέρεκ είναι να είμαστε ένα γραφείο στην πραγματικότητα που παράσχει τέτοιου είδους υπηρεσίες. Όπως βλέπετε εδώ ε, οργανώνουμε τις συνεδριάσεις του Δικού Συμβουλίου, των ομάδων εργασίας, όπως είπε ο κ. Γκότφρι, υπάρχουν εκατοντάδες εμπειρογνώμονες στους καταλόγους μας, οι οποίοι εργάζονται στα διάφορες ομάδες. Ε, υπάρχει και ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος ε, σε αυτό το μίνι συμβούλιο. Ε, εμείς υποστηρίζουμε την οργάνωση, βοηθούμε στην οργάνωση των συναντήσεων. Παίζουμε ένα ρόλο επίσης στις αναλύσεις αγοράς στις περιπτώσεις φάσης 2, από εκεί προκύπτουν κατά τις γραμμές, ε, οπότε είναι μια σημαντική διαδικασία και στα πλαίσια του κώδικα και στα πλαίσια του Μπέρεκ γενικότερα. Είναι βασικό στοιχείο δηλαδή η υποστήριξη του Μπέρεκ και επίσης υπάρχει το θέμα της διαφάνειας ε, σε ό,τι αφορά την συμμετοχή και των εμπλεκομένων φορέων, ε, των διαφορών οργανώσεων και εκεί εμείς υποστηρίζουμε αυτή την προσπάθεια. Τα τελευταία χρόνια είχαμε, όλοι, ήμασταν όλο και πιο φιλόδοξοι. Μα ζητήθηκε ε, μια πιο προωθημένη στήριξη ε, στον Μπέρε και στι εθνικέ ρυθμιστικές αρχές. Ε, συμμετέχουμε στο benchmarking, στη δημόσια διαβούλευση και τις σχετικές εκθέσεις που προκύπτουν. οργανώνουμε κατάρτιση σε ρυθμιστικό επίπεδο για, τα, για το προσωπικό. Εξετάζουμε τα ζητήματα προμηθειών, ε, μεσομελετών ε, και επίσης υπάρχει το εργαλείο ε, μέτρησης του δετερότητας, αλλά ασχολούμαστε και με τις νέες τεχνολογίες, ποιε είναι οι υποδομές που χρειάζονται για να έχουμε ψηφιακές συναντήσεις στο μέλλον. Αυτά υπήρχαν στην προηγούμενη εντολή. Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, με την νέα εντολή δηλαδή, έχουν προσθεθεί ε, κάποια νέα καθήκοντα από εσά, από του νομοθέτες. Τα πρώτα στοιχεία που βλέπετε εδώ έχουν να κάνουν με την ψηφιακή εποχή, βάση δεδομένων, προχωρημένα σύστημα πληροφορική για τη συνεργασία και βεβαίω το πέρασμα προς ε, ε, δεδομένα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να μπορούν να, να διαβαστούν από μηχανήματα. Έχουμε και κάποιες ιδέες για το μέλλον, ότι θα μπορούσαμε να επεξεργαζόμαστε εμπιστευτικέ πληροφορίε και ευαίσθητε πληροφορίε και θα πρέπει να δημιουργηθούν κατάλληλε υποδομέ γι' αυτό. Ε, υπάρχουν κάποια άλλη νέα στοιχεία στον κανονισμό, όπω παρουσίασε ο κ. Γκότφρεϊ. Τώρα πλέον έχουμε συμμετοχές, συμμετοχή και από τρίτες χώρες ε, και αυτό απαιτεί κάποια διοικητικέ, διαδικαστικέ προσαρμογέ ε, στον τρόπο συνεργασίας μας αλλά και στα συστήματά μας. Το άλλο στοιχείο επίσης είναι οι διακονισμοί εργασίας με άλλα όργανα της Ένωσης αλλά και διεθνή όργανα ε, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε λοιπόν διακανονισμούς ε, που ονομάζουμε μνημόνια, MOUs, με ε, ρυθμιστικά όργανα, ενώσεις η δέσμευση τώρα των εμπλεκομένων φορέων, η συμμετοχή τους ε, είναι σημαντική προτεραιότητα ε, και θα πρέπει να ενισχύσουμε τις δυνατότητες που έχουμε εμείς ε, στο γραφείο για να συμβεί αυτό. Και τελευταίο στοιχείο στο νέο κανονισμό Μπέρεκ είναι θα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία για τα νέα γραφεία, τη νέα εγκατάσταση με την με τη κυβέρνηση η χώρα που μας φιλοξενεί. Αυτά είναι τα στοιχεία που χρησιμοποιεί ε, το Μπέρεκ, ε, οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές, ε, όταν ασχολούνται όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πολύ σύντομα να σας πω ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις για το γραφείο Μπέρεκ στην πλαίσια της νέας συντολής του. Όπως βλέπετε, υπάρχει μια διτή προσέγγιση, πρέπει δηλαδή να υποστηρίξουμε τον Μπέρεκ και εδώ βεβαίω η πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι πρέπει να, να αναπτύξουμε τι νέε δυνατότητε και τι νέε γνώσει για να μπορέσουμε να, έχουμε, να προσφέρουμε τη μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη. Ω Μπέρεκ πρέπει να το κάνουμε αυτό ω Ευρωπαϊκή Υπηρεσία όμω. Πρέπει δηλαδή να συμμορφωθούμε με όλα τα. Ε, τους κανόνες περί κοινών ασφαλείας, προστασία προσωπικών δεδομένων, προσωπικό χρηματοδότηση, ε, την διαχείριση του κινδύνου, το μετριασμό, όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Thank uh, Σας ευχαριστώ. Καλημέρα και από μένα. Ονομάζομαι Ντόν Σρόμπλομ. Είμαι επικεφαλής του Σουηδικού EPTS ε, και ο επόμενος πρόεδρος του ΜΠΕΡΚ για το 2020. Οπότε είναι σπουδαία ευκαιρία ε, σήμερα να έρθω σε επαφή μαζί σας. Καθώς εσείς ε, φτιάχνετε την, το νέο σας, τη νέα σας εντολή Ως επερχόμενος πρόεδρος του ΠΕΡΕΚ θα έχω τη χαρά να ετοιμάσω το επόμενο πρόγραμμα εργασίας, ε, ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για τον ΠΕΡΕΚ και βεβαίως αυτό που φροντίσαμε να κάνουμε είναι ότι γνωρίζουμε πως είναι νέο το Κοινοβούλιο και ελπίζουμε πως σύντομα θα έχουμε και Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις ε, και στα δύο ε, νομοθετικά όργανα. Ωστόσο, Σήμερα δεν θα μιλήσουμε και για την επόμενη πενταετία, αλλά για το πού βρισκόμαστε στην εφαρμογή του κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών που υιοθετήσατε εσείς ως συνομοθέτης ε, ε, όχι και τόσο καιρό ε, πριν. Έχουμε το ΠΕΡΕΚ, την ευθύνη, την οποία περήφανα αναλαμβάνουμε και προσπαθούμε να φέρουμε όσο γίνεται καλύτερα εις πέρας. Έχουμε 11 κατευθυντήριες γραμμές, τις οποίες πρέπει εμείς να αποδώσουμε για μια, σε μια διετή περίοδο βασικά ξεκινώντας φέτος και τελειώνοντας του χρόνου. Τα περισσότερα πράγματα που κάνουμε είναι η επικοινωνία, κριτήρια συνεπένδυσης, επενδύσεις σε δίκτυα κτλ. Και όλα αυτά σημαίνουν ότι όπως σας είπε και ο Τζέρεμι προηγουμένως έχουμε ομάδες εργασίες οι οποίες ασχολούνται με την υλοποίηση αυτών των 11 κατευθυντηρίων γραμμών. Προτεραιότητά μας για το 19 και για το 20 είναι να ολοκληρώσουμε αυτή την εργασία με την καλύτερη δυνατή ποιότητα. Το χρονοδιάγραμμα είναι τέτοιο ώστε να φτιάξουμε την τελευταία ε, ε, τέτοια κατευθυντήρια γραμμή ε, για φέτος. Τρεις έχουμε ολοκληρώσει φέτος και του χρόνου θα μας μένουν άλλες οκτώ. Οπότε καταλαβαίνετε πως το πρόγραμμα για την επόμενη χρονιά θα είναι αρκετά αφορτωμένο. Και Τώρα θα μιλήσω για την περιαγωγή. Ξέρετε πως το Μπέρεκ έχει μακρά ιστορία στην εργασία με το, ε, για το διεθνές, τη διεθνή περιαγωγή. Είναι προτεραιότητα την οποία εξακολουθούμε να παρακολουθούμε. Παρακολουθούμε την αγορά, εκπονούμε ε, εκθέσεις σύγκριση, έχουμε εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση του κανονισμού και την εφαρμογή του κανονισμού περιαγωγής. Ε, παρέχουμε στην Κομισιόν πληροφορίες για τις νομοθετικές της προτάσεις και έχουμε ε, ε, ε, εργασίες που είναι υπό εξέλιξη αυτή τη στιγμή για την εξασφάλιση της, της ορθής εκτέλεσης του κανονισμού για την περιεχογή. Είναι όμως σημαντικό να γνωρίζουμε ότι όταν ε, καταρχάς υιοθετήθηκε αυτή, αυτός ο κανονισμός ε, για την περιαγωγή ε, υπήρχαν αμφιβολίες, όμως είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο δημοφιλή νομοθετήματα επί των οποίων εργαζόμαστε στο Μπέρεκ. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε από την αντίληψη των καταναλωτών και είχε μεγάλο αντίκτυπο στην περαιτέρω ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Καθιστά ευκολότερη τη διάβαση των συνόρων ε, τη σήμερα ημέρα, όταν ε, όλοι μας είμαστε τόσο πολύ προσκολλημένοι σε ψηφιακές μας συσκευέ. Πριν από λίγο καιρό λοιπόν ε, εισήχθη, ήταν τον Ιούνιο του 2017, μπορεί να φαίνεται πολύ χρόνος, αλλά είναι μόλις δύο χρόνια. Και όλοι βέβαια θα θυμάστε τι κάναμε όταν περνούσαμε τα σύνορα, ακόμα και μέσα στην Ένωση, πριν από αυτή την ημερομηνία, πολλοί από εμά σβήναμε τα κινητά, σβήναμε την περιαγωγή καθώς μπαίναμε στις γειτονικές χώρες και φαίνεται πως αυτή η διαδικασία σχεδόν πια έχει εξαφανιστεί. Δεν χρειάζεται να γίνεται πλέον. Βλέπουμε δε πως η κατανάλωση των υπηρεσιών ε, ίντερνετ σε άλλες ε, δικαιοδοσίες εκεί από αυτήν που έχουμε την ε, συνδρομή μας έχει αυξηθεί πάρα πολύ και αυτό βεβαίως δημιουργεί μεγάλες ευκαιρίες στην εσωτερική αγορά. Βεβαίως παρακολουθούμε όχι μόνο τα νούμερα αλλά και την εμπειρία. Ε, υπήρξαν κάποιοι αρχικοί φόβοι ότι η ποιότητα της υπηρεσίας μπορεί να μειωνόταν, ότι μπορεί να επηρεαζόταν ε, η εθνική τιμολόγηση ή η τιμολόγηση για τον υπόλοιπο κόσμο. Εμείς πιστεύουμε πως ήταν αρκετά επιτυχής η απόπειρα αυτή. γιατί μπήκαμε σε θετικό τρόπο, μπήκαμε σε θετικό τρόπο να ε, λειτουργούμε. Υπάρχουν βέβαια κάποιες ανησυχίες ακόμα, αλλά... Ε, προετοιμάζεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πιθανή αναθεώρηση του κανονισμού αυτού. Υπάρχουν επίσης κάποιες διαφορές όσον αφορά την ταχύτητα του ίντερνετ. Υπάρχει και κάποιες φορές ε, η κατάχρηση της περιεχογής. Πάντα κάποιος προσπαθεί να κερδίσει παραπάνω. Και πρέπει όλα αυτά να τα προσέχουμε. Πάντως εν γέννη ήταν μεγάλη επιτυχία. Εδώ έχετε ένα γράφημα ε, που αφορά την κατανάλωση στοιχείων. Επίση, άλλη διαφάνεια εδώ, άλλο ένα γράφημα όπου δείχνουμε με διαφορετικό τρόπο πάνω κάτω το ίδιο πράγμα. Οπότε τέλος θα ήθελα να πω κάποια πράγματα για το τι κάνει ε, το Μπέρεκ όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια. Ε, ο τομέας αυτός, όπως ε, σίγουρα θα γνωρίζετε, αναπτύσσεται ταχύτατα. Είναι ο τομέας όπου έχουμε αναπτυχθεί περισσότερο, όπου προσπαθούμε να δούμε ε, πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα και στόχος του Μπέρεκ είναι βεβαίως να μην ζητήσουμε νέα εντολή και να επικαλύψουμε την εντολή ή το ρόλο οποιοδήποτε άλλου οργανισμού ή ομάδας. Ξέρουμε πως υπάρχουν ε, άλλες ε, ε, ενδιαφέροντες οργανισμοί όπου κάνουν ε, δουλειά για την κυβερνοασφάλεια. Εμείς θα πρέπει να συνεργαστούμε μαζί τους και όχι να ανταγωνιστούμε μαζί τους. Ε, προσπαθούμε λοιπόν να αναζητούμε τη συνεργασία Φέτος ε, για πρώτη φορά έχουμε σχηματίσει ένα, μια ομάδα εργασίας με άλλες εθνικές ε, μονάδες για να εξετάσουμε τον τομέα της κυβερνοασφάλειας, για να δούμε ποιο ακριβώς ρόλο θα μπορούσαμε εμείς να παίξουμε και με τι θα μπορούσαμε να συνεισφέρουμε και να συνεργαστούμε με άλλες ομάδες, είτε είναι ε, η ομάδα συνεργασίας ΕΜΑΙΕΣ, είτε είναι η ΕΝΙΖΑ, πώς μπορούμε δηλαδή να βοηθήσουμε και να προσφέρουμε. Γνωρίζουμε ότι το 5G θα φέρει πολλούς νέους χρήστες. Πώς μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε. Είναι κάτι που ανέφερε και ο Τζέρεμι στην εισαγωγή του. Γνωρίζουμε τις αγορές πολύ καλά, γνωρίζουμε τους φορείς, ξέρουμε τι σημαίνει να ε, δουλεύει κανείς σε αυτό το τομέα. Μπορούμε δηλαδή στην ουσία να λειτουργήσουμε ως ένα συνδετικό κρίκος, μια πλατφόρμα που μπορούμε, μπορούν να συναντηθούν οι, ε, ο νομοθέτης ή ε, οργανισμοί ασφάλειας, ώστε να κινηθούμε με τέτοιο τρόπο που οι ομάδες αυτές ε, ε, ε, διαφερόντων να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή και να συνεργαστούν. Αυτό μπορούμε να κάνουμε και να προσφέρουμε με χαρά θα το κάνουμε. Έχουμε μια ομάδα εργασίας για την κυβερνοασφάλεια και φυσικά αυτή η ομάδα θα εξετάσει τι προκύπτει από την προσπάθεια της εργαλειοθήκης που κάνει τώρα η Επιτροπή να δείξουμε ότι υπάρχει βελτίωση να δούμε τι υπάρχει στην εργαλειοθήκη και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε να συμπληρώσουμε αυτή την προσπάθεια όλοι μαζί και να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια με συστήματα που να λειτουργούν ε, για όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ να προχωρήσω από το 5G και την κυβερνοασφάλεια να σας κάνω μια γενικότερη ενημέρωση για το που βρισκόμαστε με το 5G. Είναι ένα τομέας όπου το BEREC και η Κομισιόν ε, εργαζόμαστε, συνεργαζόμαστε πολύ στενά. Να σας πω τι γίνεται με την ανάθεση του φάσματος. Πριν από κάποια χρόνια είχαμε ε, εντοπίσει ότι θα υπήρχαν ε, τρεις ομάδες, μία χαμηλή στα 700 MHz, μία μεσαία ε, γύρω στα 300 MHz και μια υψηλή ε, για τους υπόλοιπους, ώστε να μπορούμε να καλύπτουμε ε, πόλεις, προάστια και αστικές περιοχές γενικά με την χαμηλή συχνότητα ε, και η ψηλότερη συχνότητα είναι για τα μέρη που υπάρχει μεγάλη πυκνότητα ζήτησης. με τις, ε, τα 700 MHz τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν ε, ξεκινήσει τις διαβουλεύσεις για να ξεκινήσουν την ανάθεση αυτών των φασμάτων ένα τέταρτο των κρατών μελών ε, το συζητάνε και τα δύο τρίτα των κρατών μελών αναμένουν την ανάθεση μέχρι τα τέλη του 2020. Τα πράγματα προχωρούν λίγο πιο αργά όσον αφορά τη 26 ε, MHz, γιατί ακριβώς η χρήση και η δυνατότητα χρήσης είναι ε, έτσι πολύ προκαταρκτική. Όλα ένα και περισσότερα κάτι μέλη ξεκινούν να καλούν τους βιομηχανικούς χρήστες που έχουν εφαρμογές να έρθουν και να συνομιλήσουν με τους ρυθμιστές ή τους ε, διαχειριστές του φάσματος για το πώς ας πούμε τα 26 GHz μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε λιμάνια ή σε μεγάλες βιομηχανίες ε, υπάρχει δηλαδή φάσμα διαθέσιμο στα 26 GHz και εν γέννη πιστεύουν όλοι ότι οι άδειε στα 26 GHz μπορεί να μην εθνικοποιηθεί όπως έχει γίνει για τις χαμηλότερες, τα χαμηλότερα φάσματα. Το σκεφτόμαστε λοιπόν για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα από άποψη χρήση. Τώρα όσον αφορά τις εμπορικές εξελίξεις, τώρα έχουμε πέντε ενάρξεις σε οχτώ κράτη-μέλη, οχτώ μάλλον, και αρχίζει να επιτεχύνεται ο αριθμός των ενάρξεων, αλλά βέβαια το ξεκίνημα είναι αργό γιατί οι συσκευές δεν υπάρχουν ακόμα. Ακόμα δεν υπάρχουν λοιπόν οι συσκευέ για το 5G, αλλά νομίζω πέρσι στη μια μεγάλη εμπορική έκθεση στη Βαρκελόνη είδαμε τέτοια πρωτότυπα. Φαντάζομαι πως του χρόνου θα είναι ακόμα περισσότερα τα κινητά ε, πέμπτης γενιάς και θα μπορούν έτσι να είναι, να, να είναι και πιο φθηνά, πιο προσιτά. ανάπτυξη της πόλης με ταχύτερη ε, ευρεία ζώνη, αλλά ακόμα και, και εκεί η χρήση των δεδομένων έχει αυξηθεί κατά τέσσερις επί τέσσερα την είδα περίοδο. Όχι τόσο γρήγορα όσο η περιαγωγή, αλλά αυξάνεται πάρα πολύ γρήγορα. Υπάρχει δηλαδή χώρος για τους ε, φορείς της κινητής τηλεφωνίας να συνεχίσουν να επενδύουν και πολύ σύντομα θα φανεί πως το 5G είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος από άποψη κόστους για την ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών. Τεχνολογία επίσης 5G για τις σταθερές ε, ε, ασύρματες συνδέσεις, ας πούμε ραδιόφωνο ε, ε, βριζονικό. Υπάρχουν πολλές δε εφαρμογές, ε, φύσεις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στις πόλεις, αλλά αυτές δεν είναι έτοιμες ακόμα για την πέμπτη γενεά. Είναι ακόμα πολύ νωρίς. Βλέπουμε λοιπόν ότι το ίντερνετ των πραγμάτων εργάζεται με βάση το 4G και με το MBIOT, όπως αυτό ονομάζεται, που είναι μια στενή ζώνη, όχι ευρεία ζώνη. Όλες αυτές οι βιομηχανικές εφαρμογές ίσως ε, να γίνουν στο 5G, αλλά μπορεί να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν και άλλου είδους εφαρμογές. Πολλές εφαρμογές δεν εξαρτώνται όμως από το 5G. Τώρα, η εργασία του Μπέριξ σε αυτό το τομέα πια είναι. Έχουμε κάνει διάφορες μελέτες τα τελευταία δύο χρόνια για επιχειρησιακά μοντέλα, για την πέμπτη γενεά, μια μελέτη για την ε, κοινή χρήση υποδομών και αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή είναι μια εργασία για το πώς θα διευκολύνουμε την καινοτομία στο 5G και στο οικοσύστημα του 5G. Δηλαδή, η ανάθεση του φάσματος είναι απαραίτητη για το 5G, αλλά μπορεί να μην αρκεί. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα ενός ζητήματος που προβλέπουμε ότι μπορεί να γίνει σημαντικό, είναι η περιαγωγή. Δηλαδή, πήρε πολύ καιρό να φτιάξουμε το κανονισμό περιαγωγής για να λειτουργήσει αυτό σωστά για το 2G, 3G, 4G, αλλά όταν ερχόμαστε στο 5G, τότε ε, ο κόσμος μιλά για μερίδες του δικτύου. Δηλαδή είναι ένας τρόπος χρήσης ε, του δικτύου 5G ώστε να προσφέρονται διάφορες υπηρεσίες ε, δεδομένων με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή ένα κομμάτι μπορεί να παρέχει μια πολύ γρήγορη υπηρεσία, ένα άλλο κομμάτι μπορεί να δίνει μια υπηρεσία με τρόπο που να λειτουργεί με συσκευές χαμηλής απορρόφησης ε, ενέργειας Άρα λοιπόν εκεί μπορεί να υπάρχει περιαγωγή ανάμεσα στα διάφορα κομμάτια του 5G και οι κανόνες που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν το εξασφαλίζουν αυτό. Γι' αυτό θα θέλαμε να μπορέσουμε να εντοπίσουμε ποιοι είναι οι, πιθαν... ποιοι... Ποιοι είναι οι πιθανοί φραγμοί που μπορεί να δημιουργούνται λόγω του ισχύοντο κανονισμού και που μπορεί να εμποδίσουν ε, αυτού του τύπου την καινοτομία. Ε, αυτό θα πρέπει λοιπόν να εντοπιστεί νωρί ώστε το Μπέρεκ να μπορέσει να δράσει ή να ε, συμβουλέψει τους αρμόδιους για την πολιτική να ενεργήσουν πριν αυτό να αποτελέσει εμπόδιο για την καινοτομία. Έχουμε ακούσει 40 διαφορετικές απαντήσεις για αυτά τα θέματα. Ε, συνήθως έχουμε μικρό αριθμό ε, σωμάτων που αντιδρούν στα ερωτηματολογιά μας, ενώ εδώ είχαμε ε, μεγάλη συμμετοχή από πλευρά της βιομηχανίας. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά έχω να σας μιλήσω ακόμα και Θα μιλήσω λιγάκι και για το ανοιχτό ίντερνετ, το οποίο είναι ε, άλλη μια νομοθεσία η οποία υιοθετήθηκε πριν από μερικά χρόνια. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ ε, νωρίς ε, ακόμα να αναθεωρήσουμε τον κανονισμό, όμως η Επιτροπή το αποφάσισε και θα πρέπει να συζητήσουμε ορισμένα θέματα σχετικά με τις κατευθυντήριες αφενός τα ενδιαφερόμενα μέρη ανησυχούσαν σχετικά με τις ε, συνέπειες που θα έχει στο 5G. Ε, είναι κάτι το οποίο το ε, διευκρινίσαμε και σχετικά με τα προγράμματα Zero Rating. Τώρα, όσον αφορά την, το κατά πόσο η Ευρώπη είναι έτοιμη για την ψηφιακή εποχή. Ε, κανείς ε, δεν ε, λέει ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουμε την νομοθεσία. Θα εφαρμοστεί στα τέλη της επόμενης χρονιάς, όμως, επόμενης χρονιάς όμως υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα ήταν χρήσιμο να εξετάσουμε ιδιαιτέρως λόγω του κόστους εφαρμογής, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τους επενδυτές στον τομέα του δικτύου της χωρητικότητας. Πιστεύουμε ότι η διαδικασία επίλυσης διαφορών ε, δεν είναι ιδιαίτερα ε, ιδιαίτερα ελκυστική και έτσι λοιπόν θα ήταν κάτι το οποίο θα, μπορούσαμε, θα μπορούσε να εξετάσει η Επιτροπή. Και επίση ε, οι κατευθυντήριε ε, σχετικά με τι κρατικέ ενισχύσει είναι 7 ε, χρονών και βασίζονται στα 30 Mbit το δευτερόλεπτο, το οποίο ήταν ο στόχο του θεματολογίου για την ψηφιακή Ευρώπη τότε και επίσης θα πρέπει να υπάρχει μια ευθυγράμμιση όσον αφορά τις διατάξεις του κώδικα. Είναι λοιπόν αυτά θέματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε και τέλος όσον αφορά ε, την ε, νομοθεσία σχετικά με την οικονομία των δεδομένων. Είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε ε, φέτο. Το ΜΠΕΡΕΚ δεν ε, προσπαθεί ε, να βρει επιπλέον δουλειά σε αυτό τον τομέα, όμω θεωρούμε ότι έχουμε πληροφορίε σχετικά με τι λεπτομέρειε τη νομοθεσία με βάση τον κανονισμό για τις τηλεπικοινωνίε. Υπάρχουν τρία βασικά θέματα, όπω είναι για παράδειγμα η, δύναμη, η αγοραία δύναμη των πλατφόρμων, η χρήση των δεδομένων των τελικών χρηστών, η Επιτροπή, τα κρατημέλη αλλά και αλλού στον πλανήτη υπάρχουν ε, αιτήσει ε, για περαιτέρω ε, νομοθέτηση σε αυτόν τον τομέα και θεωρούμε ότι από πρακτικό τομέα δεν είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο για διάφορους λόγους αφενός διότι ο ρυθμός καινοτομία σε αυτές τις πλατφόρμες είναι πάρα πολύ γρήγορο σε σχέση με το πώ λειτουργεί η νομοθετική διαδικασία και επίση έχουμε θέματα τα οποία αφορούν την εμπειρογνωμοσύνη, το συνδυασμό των, της γνώσης που υπάρχει πάνω σε αυτό και φυσικά υπάρχουν και ε, υπερεθνικές και εθνικές διαστάσεις. Θα θέλαμε λοιπόν να κάνουμε μια προσφορά ε, στους θεσμούς να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Υπήρξε μια ανάλυση της αγορίας δύναμης ε, των κανόνων εξάντε, ιδιαίτερα όσον αφορά την αγορά δύναμη. Τα δεδομένα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει μελλοντικό όπως έκανε οι υποδομές στο παρελθόν. Επίσης, ο ανταγωνισμός είναι ένα θέμα και τέλος, σίγουρα θα υπάρχει μια ανάγκη τόσο για υπερεθνικές και εθνικές ε, διαστάσεις ε, και ο Μπέρεκ παρουσιάζει παραδείγματα ε, επιτυχημένου δικτύου όπου οι νομοθέτες από διάφορα κράτη-μέλη μπόρεσαν να θεσπίσουν ένα κοινό νομοθετικό πλαίσιο. Και θα σταματήσω τώρα εδώ και θα δώσω το λόγο πάλι στον ε, πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Godfrey, για την εισαγωγή σας και έχουμε έναν πρώτο γύρο ερωτήσεων. Θα ξεκινήσουμε αμέσως ε, με την κυρία Καβαλιού. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή σχετικά με το ρόλο του ε, Μπέρεκ ε, και τις υπηρεσίες που τον υποστηρίζει. Όντως ε, μπορούμε να κάνουμε πολλά σχετικά με την ψηφιακή ολοκλήρωση της αγοράς και τις ηλεκτρονικές τηλεπικοινωνίες. Θα ήθελα να θέσω τρεις ερωτήσεις τώρα υπήρξε ένας, ε, μια διαφάνεια σχετικά με το 5G. Όμως ε, ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος ε, του Μπέρεκ ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα μείνουν πίσω κάποια κράτη-μέλη κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. ότι θα αναπτυχθούν οι απαραίτητε διαδικασίε ε, και τεχνολογίε που θα μα προετοιμάσουν ε, για το μέλλον όσον αφορά το διαδίκτυο των πραγμάτων και το 5G. Ε, θα μπορούσατε να αναλάβετε τον ρόλο για την ανταλλαγή πληροφοριών για να προωθήσετε τα κράτη-μέλη. Το δεύτερο ερώτημα τώρα είναι ότι θα θέλατε να συμμετάσχετε σε αυτή την οικονομία δεδομένων. Όμως δεν θέλετε να αναλάβετε κεντρικό ρόλο πάνω σε αυτό. Είπε κάποιος από εσά στην αρχή ότι θα είναι σημαντικό ε, να ε, ε, να, να υπάρχουν τα δεδομένα σε μια τέτοια μορφή ώστε να μπορούν να είναι αναγνώσιμα από μηχανές. Όμως αυτό δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν διάφορα δεδομένα τα οποία όμως δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο εύκολα, δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε τόσο εύκολα, ε, γιατί δεν επαναχρησιμοποιούνται. Οπότε, τι ρόλο μπορείτε να παίξετε ε, πάνω σε αυτό, ώστε να δημιουργηθούν αυτά τα πρότυπα, ούτως ώστε πραγματικά τα δεδομένα να μπορούν να χρησιμοποιούνται. Και τέλος, όσον αφορά τους καταναλωτές αναφέρατε τους ε, καταναλωτές στο πλαίσιο της περιαγωγής. Όμως ε, ε, οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες είναι ένας τομέας όπου οι καταναλωτές διαμαρτύρονται περισσότερο. Τι κάνετε λοιπόν, ούτω ώστε ε, να υπάρχουν οι βέλτιστες πρακτικές, ούτω ώστε οι ε, καταναλωτές να βρίσκονται στο επίκεντρο των ε, στρατηγικών των εταιριών και των κρατών μελών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Καβάλιο και τώρα από τους σοσιαλιστές ο κύριος Νικά. Ευχαριστώ πολύ. Έχω μία ερώτηση ε, σχετικά με την όλη διαδικασία. Αρχικά, ισχύει ότι η Επιτροπή έχει ως στόχο της να παρουσιάσει μία ανακοίνωση και θέλει να παρουσιάσει τις κατευθυντήριες για τους παρόχους για να ε, διασφαλίσει ότι ε, τα κράτη-μέλη κατά τη διάρκεια των ε, διαγωνισμών θα έρχουν μια μεγαλύτερη προσέγγιση όσον αφορά την ανεξαρτησία των παρόχων και σε περίπτωση που κάτι τέτοιο ισχύει, ποια είναι η θέση σας πάνω στο θέμα αυτό. Έρχομαι από την Ρουμανία και ε, πρόσφατα όπως ότι η ρυθμιστική αρχή της ε, Ρουμανίας ε, ήθελε να, αναβάλει τον διαγωνισμό μέχρι ότου να υπάρχει ένα μνημόνιο συμφωνίας συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου θα αναγνωρίζονται οι συνθήκες για τους παρόχους και θα είμαστε πιο επιλεκτικοί ε, σχετικά με το ε, ποιοι ε, πάροχοι 5G θα επιλέγονται. Βλέπω ότι υπάρχουν διάφορες απόψεις στα κράτη-μέλη και γνωρίζω ότι ο Μπέρεκ προσπάθησε να υπάρξει μια ενιαία προσέγγιση σε, όλες σε όλα τα κομμάτια της διαδικασίας Πώς ε, θα απαντούσατε λοιπόν αυτό το θέμα. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να εισάγουμε αυτές τις ε, νέες συνθήκες ε, και να υπάρχει μια ίση μεταχείριση όλων των κρατών μελών, να έχουν μια κοινή, μεταχείρι... μια κοινή προσέγγιση, ένα κοινό όραμα, διότι υπάρχει η τάση να, όπου ε, θα έχουμε μια προσέγγιση για όλα τα κράτη-μέλη στο σύνολό τους. Θα μπορούσατε λοιπόν να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες ε, για αυτό, διότι ε, μας λείπουν οι ε, σωστές απαντήσεις πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ κύριε Νίκη. Από τους πράσινους ο κύριος ε, Νινίστο, ευχαριστώ ε, πολύ ε, για, την, ε, παρουσία, για τις παρουσιάσεις σας. έχω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την περιαγωγή. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία και είναι κάτι το οποίο εκτιμούν ιδιαίτερως οι καταναλωτές. Όμως υπάρχουν και κάποιες ανησυχίες Ορισμένοι πάροχοι έχουν αυξήσει ε, τις τιμές τους ε, ε, σε εθνικό επίπεδο για να μπορέσουν να καλύψουν τα έξοδά τους στο εξωτερικό. Και έτσι δεν έχουμε επικεντρωθεί στο ζήτημα του κόστους στην νομοθεσία. Ήταν λοιπόν ε, μια παραπέμπτωση συνέπεια σε ορισμένα κρατημέλη. Ένα άλλο ερώτημα τώρα σχετικά με την παραγωγή επίση. Πώς μπορούμε να το επεκτείνουμε, είναι κάτι το οποίο, τι μπορούμε να κάνουμε ε, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τόσο ώστε να επεκτείνουμε την διαθεσιμότητα αυτές της ε, υπηρεσίας. Ευχαριστώ πολύ. Από το ECR, ο κύριος ε, ε του Σουνόφσκι, όπου ήταν και εισηγητής ε, γνωμοδότηση πάνω σε αυτό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εισαγωγή των ε, δραστηριοτήτων ε, του Μπέρεκ ε, και τις υπηρεσίες που υποστηρίζουν τον Μπέρεκ. Κατανοώ ότι ε, δεν είναι εύκολο να ε, κατανοήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Κατανοώ ότι σίγουρα θα υπάρχουν πολλοί και εδώ στο Κοινοβούλιο που θα αντιμετωπίζουν δυσκολίες ε, με την κατανοήση σχετικά με το πώς συνεργάζονται οι διάφορες τεχνικές αρχές με τον ΠΕΡΕΚ και γι' αυτό το λόγο ευχαριστούμε που διοργανώσατε αυτή την ενημέρωση εισηγητής της γνωμοδότησης για το θέμα αυτό πέρσι. Ήμασταν σε επαφή για αρκετούς ε, μήνες ε, και ευχαριστώ ε, που καταφέραμε να διαχειριστούμε το θέμα σχετικά με τον κώδικα Τώρα, το πρώτο θέμα για τους νομοθέτες όσον αφορά την εφαρμογή του κώδικα ε, θα ε, θέλαμε ο ε, μελλοντικός πρόεδρος του Μπέρεκ να μας ενημερώσει ποιες ε, θα είναι οι μελλοντικές προκλήσεις. κατανοήσαμε πόσο πολύπλοκη θα είναι η διαδικασία εφαρμογής. Τώρα το δεύτερο ερώτημα αυτό το οποίο βλέπουμε ε, και ε, σε άλλα κράτη-μέλη ε, είναι ότι υπάρχει υποχρηματοδότηση του Μπάρακ. Θα πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση, να αυξηθεί το προσωπικό, όπως είπατε και οι ίδιοι. Οι προσδοκίες και οι απαιτήσει που υπάρχουν για τον Μπέρεκ θα αυξηθούν. Έτσι λοιπόν, τι πρόοδο βλέπετε σε αυτό το ε, θέμα. Αυτό το οποίο θα ήθελα ε, να ακούσω λοιπόν είναι ποια είναι τα επιχειρήματα για την ενίσχυση ε, του Μπέρεκ και τρίτον στον κανονισμό για τον Μπέρεκ υπάρχει η δυνατότητα απασχόλησης ε, του προσωπικού του Μπέρεκ εκτός ε, των ε, γραφείων του Μπέρεκ σε μια άλλη πόλη ούτως ώστε να υπάρχει μια στενότερη επαφή με τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Ποια η θέση σας για το θέμα της ε, δημιουργίας ενός ε, μικρού ε, γραφείου σε μια άλλη πόλη. Και για τον συνάδελφό σας κύριο Νιέτσι αναφερθήκατε ε, στην ε, συμφωνία με την ε, κυβέρνηση της Λετωνίας ποιο είναι το χρονικό πλαίσιο και τι πιστεύετε ότι θα ήταν αναγκαίο ούτως ώστε να αναθεωρήσουμε τη συγκεκριμένη συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τωσενάφσκι, αυτός ήταν ο πρώτος γύρος των συντονιστών. Ελπίζω να μπορείτε να χωρίσετε τις ερωτήσεις μεταξύ σας και να δώσετε κάποιες απαντήσεις με κάποια σειρά. Ναι, ευχαριστώ. Μοιράζουμε εμείς τις απαντήσεις. Να απαντήσω πρώτα στην κυρία Καρβάλιο. Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη θα μείνουν πίσω σε ό,τι αφορά το 5G. Ένα από τα ζητήματα έχει να κάνει βεβαίως με την διάθεση του φάσματος. Ε, υπάρχει, υπάρχουν προβλήματα ε, συνεργασίας με κάποιες ε, συνοριακές ε, χώρες που δεν είναι κρατημέλη, ιδιαίτερα στα ανατολικά μας σύνορα, κάποια κρατημέλη δημιουργούν προβλήματα που δεν έχουν άλλα κρατημέλη. Και εκεί χρειάζεται κάποια αμοιβαία συνδρομή, ε, ανταλλαγή εμπειριών. Εγώ θα έλεγα το λέτε και ότι στον κώδικα υπάρχει μια διάταξη για αξιολόγηση ομοτήμων σε ό,τι αφορά αυτές τις διαδικασίες. Δεν έχει ακόμα βέβαια ε, εφαρμοστεί, όπως και να έχει πάντως. Έχουμε κάποιους ε, διακονισμούς εργασίας μεταξύ μας και έχουμε τακτικά οργανώνουμε εργαστήρια με διαχειριστές φάσματος ε, και άλλους με άλλα μέλη του Μπέρεκ για να ανταλλάξουμε πληροφορίες ε, για ορισμένα επιμέρους ζητήματα. Είχαμε ένα εργαστήριο πριν από μία ή δύο εβδομάδες όταν και συζητήσαμε κάποια από τα θέματα ε, του τι γίνεται με τα 26 GHz, ε, τι γίνεται με τις ανησυχίες για την υγεία που έχουν εκφράσει κάποιοι, πώς μπορούμε να καθησυχάσουμε το κοινό για τις ε, επιπτώσεις για την υγεία του των, από τα 5 από το 5G. Έχουμε λοιπόν ανταλλαγή εμπειριών. Ε, τώρα για τη χρήση ε, κάποιοι πιστεύουν, κάποιοι στον Μπέρεκ είναι μια προσπάθεια μάλλον να εξασφαλίσουμε ότι όταν έχουμε μια πανευρωπαϊκή ένα πάροχο πανευρωπαϊκών υπηρεσιών, μια startup παραδείγματο χάρη που θέλει να αναπτύξει ένα ίντερνετ των πραγμάτων ανά την Ευρώπη, ε, προσπαθούμε να εντοπίσουμε ποια είναι τα θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε έτσι ώστε να μπορεί να γίνει αυτό όσο γίνεται λιγότερε τριβέ. Τα κάνουμε αυτά λοιπόν. Μα ρωτήσατε και για τα επαναχρησιμοποιούμενα δεδομένα. Εδώ υπάρχουν δύο πτυχέ. Πρώτον, τα δεδομένα του Μπέρεκ, του ίδιου του Μπέρεκ δηλαδή, ε, εξετάζουμε πώς μπορούμε αυτά τα δεδομένα να είναι πιο εύκολα διαθέσιμα έτσι ώστε όταν ε, δημοσιεύουμε την έκθεσή μας για την περιαγωγή για άλλα πράγματα που συμβαίνουν στην αγορά ε, με τον καιρό προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό ηλεκτρονικά ε, ή να μπορούμε να το κατεβάσει κάποιος να το φορτώσει ηλεκτρονικά ε, υπάρχει ένα ευρύτερο θέμα με την ψηφιακή οικονομία που έχει να κάνει με τις μεγάλες πλατφόρμες ε, και πώς θα μπορούν τα δεδομένα να είναι φορητά ε, πώς θα μπορούν να είναι προσβάσιμα με τη χρήση, με την ε, με του χρήστη βέβαια. Ε, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό αυτό και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε στις συζητήσεις για τον μελλοντικό κανονισμό. Και βέβαια στα ζητήματα διαλειτουργικότητας και πρόσβασης είναι ζητήματα όπου υπάρχουν σχετικά, σχετικές αναλογίες και στον κανονισμό για τις τηλεπικοινωνίες, αλλά δεν, μπορούν, ισχύουν όμως, δεν μπορούν να ισχύσουν ακριβώς τα ίδια εδώ. Ε, επίσης ρωτήσατε για τους τελικούς χρήστες και τους καταναλωτές. Προφανώς και είναι ζωτική σημασία σε αυτό για τον Μπέρεκ. Ό,τι κάνουμε ε, για να αυξήσουμε τον ανταγωνισμό, ο ανταγωνισμός αυτός ε, τον, εμείς τον εννοούμε με τον καλό τρόπο, δηλαδή ότι μπορεί να βελτιώσει τα πράγματα για τον τελικό χρήστη, για τον καταναλωτή. Ένα από τα μέσα στις που κάνουμε είναι το Contract Summary Templates. Είναι ε, κάτι νέο που προβλέπει ο κώδικα, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι ο καταναλωτή όταν επιλέγει μεταξύ παρόχων να, έχουν πληροφο... να έχει πληροφορίε για το τι αγοράζει και αυτό να γίνεται με μια μορφή που να είναι πανομοιότυπη, να είναι συνεπής από τους διαφόρους παρόχους, να μπορούν να συγκρίνουν ε, γίνεται και μια δουλειά για την πρόσβαση ε, των ατόμων με αναπηρία σε, αυτά τα, ε, σε αυτές τις υπηρεσίες. Γίνεται μια προσπάθεια για να θεωρηθεί καθολική υπηρεσία αυτή. Θα πρέπει όλα τα κρατημέλη να εξασφαλίσουν ότι θα είναι διαθέσιμο το κατάλληλο ευρύ φάσμα σε όλους τους τελικούς, τελικούς και να δούμε τις βέλτιστες πρακτικές και πώς θα ξεχωρίσουμε καλύτερα αυτά που εννοούμε. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο έχει να, που έχει να κάνει με τους τελικούς χρήστες είναι όταν έχουμε πληροφορίες ε, σχετικά με την κάλυψη, την κινητή κάλυψη, πώς αυτή η πληροφορία θα φτάνει στον τελικό χρήστη, πώς θα γνωρίζει ο, ο πότε έχει καλή κάλυψη, πότε έχει μοριακή κάλυψη, διότι οι πληροφορίες για την κάλυψη που δίνουν, που δίνουν οι η παροχή είναι ας πούμε αισιόδοξοι, έτσι. Ε, και έχουμε κάνει λοιπόν κάποια δουλειά εμείς ως Μπέρεκ ε, και μια σειρά από αρχές ε, σε κράτη-μέλη έχουν βοηθηθεί από τη δουλειά που έχουμε κάνει. Ε, να απαντήσω σε κάποια από τα ερωτήματα του κ. και στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Ο κ. θα θέσατε ένα ερώτημα για το γραφεία του Μπέρεκ, το γραφείο του Μπέρεκ, τον προπολογισμό του και το προσωπικό. Ε, το Μπέρεκ πέρυσι, ίσως και νωρίτερα, είχε πει ότι το προσωπικό πρέπει να αυξηθεί του γραφείου του Μπέρεκ, ε, διότι όπως ελέγχθη, το γραφείο του Μπέρεκ είναι η πιο μικρή υπηρεσία της Ένωσης. Και ένα από τα προβλήματα για μια μικρή υπηρεσία είναι ότι χρειάζεται ένα ελάχιστο αριθμό προσωπικού για να συμμορφωθούμε με τους κανόνες ε, διοίκησης, οικονομικής διοίκησης. Υπάρχει ο κίνδυνος λοιπόν ότι ε, οι άνθρωποι αυτοί να ασχολούνται τελικά με τα διοικητικά και να μην κάνουν πραγματική δουλειά για την οποία υπάρχει υπηρεσία. Είναι ένα ζήτημα που το γνωρίζουμε, ε, το έχουμε συνειδητοποιήσει και είχαμε προτείνει νομίζω 12 ή 14, προτείναμε 14 άτομα ε, δύο λάβαμε τον προπολογισμό. Ε, σε ό,τι αφορά τα ε, χρήματα, ε, έχουμε καταφέρει να έχουμε συμβασιούχους και εθνικούς εμπειρογνώμονες για να κάνουν τη δουλειά του γραφείου του Μπέρεκ. Δεν είναι όμως και τόσο ικανοποιητικό το αποτέλεσμα, διότι τελικά όταν δεν έχουμε μόνιμο προσωπικό, ψάχνουμε πολύ περισσότερους ανθρώπους ε, έχει κάποιες εργασίες δεν μπορούν να τις κάνουν οι ίδιοι άνθρωποι. Ε, θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια προσπάθεια ε, για να έχουμε περισσότερο μόνιμο προσωπικό και λιγότερους συμβασιούχους. Ε, τα κράτη-μέλη συχνά είναι επιφυλακτικά, υπάρχουν δημοσιονομικά ζητήματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο του Διοικητικού Συμβουλίου του Μπέρεκ, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Επίσης, ρωτήσατε κατά πόσο πρέπει να υπάρχει ε, ένα γραφείο δορυφόρος κάπου στις Βρυξέλλες. Ε, έτσι πως δουλεύει το Μπέρεκ, ε, το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς γίνεται στις ομάδες εμπειρογνωμόνων, στις ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων και από, βεβαίως από το, το Συμβούλιο Ρυθμιστικών Αρχών. Και εμείς ε, το, το γραφείο του Μπέρεκ υποστηρίζει αυτές τις δουλειές. Δηλαδή πολλές συνεδριάσεις ούτως ή άλλως από χώρα στις Βρυξέλλες. Ε, εγώ ως πρόεδρος του Μπέρεκ ε, κάποια στιγμή θα πρέπει να αγοράσω ένα διαμέρισμα στις Βρυξέλλες, τόσο καιρό περνάω εδώ. Ε, δεν ε, τα πάμε και τόσο άσχημα στη σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι άλλε υπηρεσίε. Το συζήτησε αυτό το συμβούλιο του, Μπέ, του Μπέρε κατά πόσο πρέπει να υπάρχει ένα γραφείο δορυφόρο για την ώρα δεν είναι προτεραιότητα. Ε, Βεβαίω ε, το συζητούμε ε, και με τη λεπτονική κυβέρνηση για το τι θα γίνει με, με τι εγκαταστάσει μα. Θα δούμε πώ θα πάνε οι συζητήσει αυτέ και αναλόγως ε, θα δούμε εάν θα υπάρξει κάποιο γραφείο στις Βρυξέλλες. Για την ώρα πάντως δεν θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο. Ναι, για, το, για την έδρα. Να σας πω για τη σχετική συμφωνία. Ευχαριστώ το Σονόσκι για το ερώτημα, αλλά και για την υποστήριξή σας ε, κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας των διαφορών προκλήσεων που αντιμετωπίσαμε για το θέμα, στα θέματα των πόρων, λοιπόν για το χρονοδιάγραμμα σε ό,τι αφορά την έδρα. Όπως αναφέρει ο νέος κανονισμός Μπέρεκ, ε, έχουμε ε, ένα χρονικό διάστημα δύο ετών για να συμφωνήσουμε με, τη λετωνική, με, τις λετωνικές, με τις λετωνικές αρχές, ξεκινώντας από το Δεκέμβριο του 2018. Το πρώτο έτος χρησιμοποιείται για την προπαρασκευή και την αξιολόγηση. Ήδη το Συμβούλιο έχει εγκρίνει μια εντολή ε, με συγκεκριμένους στόχους Ήδη το Μάρτιο φέτος έγινε αυτό. Η λετωνική κυβέρνηση είναι στη διαδικασία ολοκλήρωσης ενό παρεμφερούς εγγράφου, το οποίο ονομάζουν έγγραφο θέσεων, όπου θα αναφέρονται οι παράμετροι, οι στόχοι για τη νέα αυτή συμφωνία. Και αυτό το έγγραφο θα είναι έτοιμο σε λίγες μέρες. Αυτή είναι η διαδικασία. Στο δεύτερο έτος θα συμφωνήσουμε για τα νέα γραφεία και όλοι θεωρούμε ότι αυτή τη φορά ε, ότι αυτός αυτό το χρονικό διάστημα θα είναι αρκετό. Ε, υπάρχει υποστήριξη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις υπηρεσίες της, ε, ιδιαίτερα από την DG Connect, για να αντιμετωπίσουμε μια σειρά από οριζόντιε προκλήσει σε ό,τι αφορά τη συμφωνία αυτή για, τα, για τι νέε καταστάσει μα. Ρωτήσατε και για το ποιοι τομείς, σε τομεί πρέπει να υπάρξει επικαιροποίηση σε αυτήν την συμφωνία. Να σα πω ότι έχουμε εντοπίσει τρία ζητήματα. Το, θέμα είναι, το, το, το ένα θέμα είναι τα ίδια τα γραφεία, τι ίδιε καταστάσει πριν από 10 χρόνια μα ε, τα είχαν χορηγήσει αυτά, οπότε κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει και μια ανανέωση. Το δεύτερο είναι το καθεστώ τη υπηρεσία. Αυτό είναι ένα ζήτημα ε, για κάθε κράτο μέλος να, να μπορέσει το πρωτόκολλο παρθμών 7 να κουμπώσει με την εθνική νομοθεσία. Υπάρχουν τα ζητήματα επιστροφή ΦΠΑ, παραδείγματο χάρη, να δώσω ένα παράδειγμα. Και το τρίτο είναι το καθεστώς ε, του προσωπικού, πάντα σύμφωνα με το πρωτοκόλλο ε, παριθμών 7, ε, το καθεστώς του προσωπικού και των μελών της οικογένειας είναι πολύ συγκεκριμένο στα κράτη-μέλη και εδώ έχουμε προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε, αλλά υπάρχει καλή βούληση, υπάρχει έτσι, επικοδομητικό πνεύμα και από τις δύο πλευρές και νομίζουμε ότι θα υπάρξει αρκετός χρόνος. και όπως μου λένε εδώ στο αυτή υπάρχει το θέμα ε, των, του Ευρωπαϊκού Σχολείου ε, που στον κανονισμό και είναι κάτι που θα πρέπει να και αυτό να επιληθεί στη νέα συμφωνία. Μάλιστα να σχολιάσω και εγώ νομίζω υπάρχουν τρία ερωτήματα που μένουν. Το ένα είναι από τον κύριο Νίκα για τις συζητήσεις σχετικά με την κυβερνοασφάλεια. Όπως θα θυμάστε την Άνοιξη υπήρξε μια σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ότι το κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν μια άσκηση αξιολόγηση κινδύνου για το μοντέλο αξιολόγηση κινδύνου και να παρουσιάσουν τις μελέτες ε, που θα κάνουν ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τη συμπτύξει και να συνεχιστεί από εκεί πέρα η συζήτηση. Εκεί βρισκόμαστε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προετοιμάσει μια έκθεση μετά από όλα αυτά και αυτή την εργαλειοθήκη στην οποία αναφέρθηκα στην αρχική μου δήλωση και εκεί συμμετέχουν πολλές εθνικές αρχές ε, σε εθνικό επίπεδο ε, κάποιοι δραστηριοποιούνται και στα πλαίσια της ΕΝΗΣΑ η ασφάλεια είναι ένα ζήτημα εθνικής αρμοδιότητας οπότε σε ό,τι αφορά την εναρμόνιση αυτό που θα συμβεί ε, θα είναι μια μαλακή εναρμόνιση που προκύπτει από την ε, ε, συζήτηση, την ενημέρωση, την αλληλοενημέρωση για τις διάφορες πολιτικές επιλογές. πολλά πράγματα γίνονται. Έγινε η διάσκεψη για την κυβερνοασφάλεια στην Πολωνία πριν από μερικές εβδομάδες. Με μεγάλη συμμετοχή από όλη την Ευρώπη τα κράτη-μέλη, τα θεσμικά όργανα και όλοι νομίζω έχουν αντιληφθεί ε, ποια είναι τα ζητήματα που προκύπτουν από την ε, εισαγωγή σε μεγάλη κλίμακα του 5G ε, και του διαδικτύου των πραγμάτων. Όλα αυτά πολλαπλασιάζουν τα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, παραλήπτες, δέκτες, εκπομπές. Θα πρέπει να υπάρχει ένα επαρκές επίπεδο ασφάλειας για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές, αυτά τα φανταστικά μηχανήματα ε, για την σωστή χρήση τους όμως. Χωρίς να δημιουργούνται κίνδυνοι αχρίαστοι σε αυτή τη διαδικασία. Δεν νομίζω ότι το Μπέρεκα θα συστήσει κάποια συστήματα ή κάποιους προμηθευτές ε, ε, αυτό που μπορούμε να κάνουμε με τους φίλους μας από άλλες οργανώσεις είναι να προωθήσουμε ευέλτιστες πρακτικές ό,τι αφορά τις διαδικασίες, ό,τι αφορά τα μοντέλα αξιολόγηση κινδύνου, ε, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση ε, των πιο ευαίσθητων ε, πλευρών του εξοπλισμού διαδικτύου, τέτοια πράγματα. Το Μπέρεκ πάντως δεν νομίζω να είναι σε θέση να ε, συστήσει πιο λεπτομερώς ε, ποιος πρέπει να είναι ο εξοπλισμός στο διαδίκτυο ούτε το Μπέρεκ ούτε τα εθνικές αρχές είχαν κάποια σαφή θέση για το ποιο εξοπλισμό πρέπει να χρησιμοποιούν ε, και πώς θα πρέπει τα δίκτυα των διαφόρων παρόχων να δομηθούν. Δεν μπορεί να το κάνουμε αυτό, διότι δεν είναι μια ευθύνη την οποία δεν μπορούμε να αναλάβουμε, να επομισθούμε. Να περάσω τώρα στο θέμα της περιαγωγής. Όπως αναφέρθηκε, σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε αναφορές ε, για αύξηση των εσωτερικών τιμών. Ε, είναι πάντα δύσκολο να ξέρει κανείς κατά πόσο αυτή η αύξηση ε, σχετίζονται με την περιαγωγή. Η σχέση αιτίας αιτιατού δεν είναι και τόσο σαφής. Είναι πάντως πολύ καλή αυτή η νομοθεσία. Εμείς παρακολουθούμε την εφαρμογή της. Θα υπάρξει μια νέα έκθεση το 2021 νομίζω. Θα το ξαναδούμε και θα δούμε και τι θα έχει γίνει και με το 5G. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε τρεις ε, συναδέλφους που έχουν να θέσουν ερωτήσεις και 12 λεπτά για να κλείσουμε αυτό το θέμα. Έχουμε χρόνο. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Κέλλη κύριος Κέλλη. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ ε, όλους σας για τις ε, παρουσιάσεις σας. Πολύ ενδιαφέρουσες. Έχω δύο ερωτήσεις. Η μία αφορά το θέμα της ε, ε δυνατότητας σύνδεσης απαιτήσει για την σύνδεση. Πού βρισκόμαστε στην Ευρώπη ως προς αυτό και εσείς τι βλέπετε, ποιος βλέπετε Πώς βλέπετε να γίνεται ε, αυτός ο, αυτή η σύνδεση σε ολόκληρη την Ευρώπη τα επόμενα δέκα χρόνια. Έπειτα η περιεγωγή ήταν επιτυχία του Μπερέκ, του Κοινοβουλίου και της Ήτρε και ειδικά για ανθρώπους όπως η Πιλάρ που αρισχολήθηκε με το θέμα αυτό για πολλά χρόνια. Ε, τώρα, για την περιεγωγή, πώς επηρεάστηκαν τα κέρδη των εταιριών τηλεπικοινωνίας. είχε προβλεφθεί πως θα υπήρχε αύξηση στη χρήση της κινητής τηλεφωνίας. Έχετε στοιχεία γι' αυτό και έπειτα τα ωφέλη ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πώς, ε, ε, ποια είναι. Ευχαριστώ κύριε Κέλλη, κυρία ε, Κομπελανίτσε. Ευχαριστώ. Υπάρχει ανάλυση, καμία ανάλυση όσον αφορά την ιδιοκτησία των δεδομένων για την προθεσμία τη περιαγωγής. Πότε πιστεύετε πως θα είστε έτοιμοι για την ανάλυση 5G, γιατί ολόκληρος ο κανονισμός θα έχει λήξει σε δυόμιση χρόνια. Είναι αργή η διαδικασία, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε και για πάρα πολύ. Έπειτα, ευρεία ζώνη για όλους. Έχετε αναλύσει την αγορά ε, του ε, και πώς ακριβώς θα γίνει αυτό. Θυμάμαι ότι για το 5G ας πούμε πώς μπορούμε να το έχουμε όπως στη Σκανδιναβία, δεν είναι όλοι έτοιμοι οι φορείς να το προσφέρουν μέσα σε λίγες μέρες το, το 5G. Και έπειτα η ερώτηση του συναδελφού Νίκα για την ε, δυσλειτουργία, την κυβερνοασφάλεια. Είναι δυνατόν το Μπέρεκ να προτείνει τουλάχιστον κάτι που να είναι γενικό για όλη δηλαδή την εσωτερική αγορά. Εγώ Καταλαβαίνω ότι θα θα μπορούσε να είναι κάτι το γενικό, εάν είναι καλό ή κακό, κάποιος μπορεί να το επιστρέψει. Είναι ψυγείο, αν είναι υπολογιστή αν είναι το δίκτυο ή κομμάτι του δικτύου. Να υπάρχει δηλαδή αυτός ο κανόνας ότι θα μπορούμε αυτό το κομμάτι να το απομονώσουμε. Να έχουμε δηλαδή έναν ελάχιστο κοινό παρονομαστή. ευχαριστώ. Κυρία Σόλης Σεμπέρε, στα Ισπανικά θα μιλήσω παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας. Εσείς ε, αναφέρατε την ανάθεση του φάσματος για βιομηχανική χρήση και ήθελα να ξέρω ποια είναι η γνώμη σας. Ξέρετε ότι το, ο γερμανικός ρυθμιστής ε, αποφάσισε ότι θα δώσει ένα κομμάτι του φάσματος για τοπικές, ε, τοπικά ραδιόφωνα. Δηλαδή δεν θα βάλει σε πληστηριασμό αυτό το κομμάτι του φάσματος αλλά το θέσει στη διάθεση της βιομηχανίας. Δεδομένης της σημασίας του 5G για το ίντερνετ πραγμάτων για τη βιομηχανία. Εσείς πιστεύετε πως τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ακολουθήσουν αυτό το μοντέλο και να δώσουν ένα κομμάτι του φάσματος για βιομηχανική χρήση, γιατί η ανάθεση του φάσματος είναι εθνική αρμοδιότητα, το ξέρω. Αλλά θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η δική σας γνώμη για το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Η κυρία Τόγια, τελευταία ερώτηση. Σας ευχαριστώ. Εγώ θα μιλήσω Ιταλικά, παρακαλώ. Βάλτε τα ακουστικά σας. Ευχαριστώ. Να εδώ κάθομαι. Θέλω πολύ πολύ σύντομα, επειδή α, άκουσα διάφορες, απαντήσεις, διάφορες ερωτήσεις για την περιεχογή, άκουσα τη δική σας απάντηση και πρέπει να σας πω πως ήταν λίγο έτσι βιαστική, ίσως λόγω χρόνου. Το δικό μου ερώτημα είναι το εξή. ως σκιώδης για την διάταξη που έφερε στην κατάργηση του εισπεραγωγής και η συγγήτρια ήταν η συνάδελφος Καρβάλιο, θα ήθελα να ζητήσω την προσοχή σας, την απόλυτη προσοχή σας, γιατί από πολιτική άποψη ήταν ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχει κάνει κάνει η Ευρώπη, λένε οι πολίτε. Οπότε πρέπει να αποφύγουμε κάθε απόπειρα να παρακαμφθεί αυτή η διάταξη με ένα σωρό ε, παράξενες ε, ε, χρεώσεις. Ας πούμε, την πρώτη μέρα έγινε απόπειρα να ερμηνευθεί διαφορετικά η χώρα της ε, διαμονής. Ε, ε, θα πρέπει λοιπόν το Μπέρεκ να προσέχει διαρκώς και απόλυτα την εφαρμογή αυτής της διάταξης που όπως είπαμε ήταν πολύ σημαντικός ε, κανονισμός για την ευρωπαϊκή πολιτική και δεν πρέπει να αφήσουμε να παρακαμφθεί ε, από διάφορες ε, επιτίδιους. Ευχαριστώ. Τώρα έχετε πέντε λεπτά για να απαντήσετε και να κλείσετε. Ξέρω πως μπορείτε να τα καταφέρετε. για τα συνδεδεμένα οχήματα. Προφανώς, το μέλλον των αυτόνομων συνδεδεμένων αυτοκινήτων είναι πολύ σημαντικό. Μια από τις απόψεις του Μπέρεκ που είχαμε για αυτά τα επιχειρηματικά μοντέλα είναι ότι δεν θα είναι μια επανάσταση στη δυνατότητα σύνδεσης. Μάλλον, αυτόνομα οχήματα πρέπει να μπορούν να λειτουργήσουν σε περιοχές που υπάρχει το 3G, το 4G αλλά και το 5G. Δηλαδή οι κατασκευαστέ αυτοκινήτου δεν θα φτιάξουν αυτοκίνητα τα οποία να μπορούν να οδηγηθούν μόνο σε περιοχέ που καλύπτονται από το 5G. Είναι σημαντικό λοιπόν να φτάσουμε στο 5G, ναι, αλλά η αυτοκινητοβιομηχανία ε, θα πρέπει να προχωρήσει ούτως ή άλλως. Υπάρχει δεν υπάρχει ε, η κάλυψη 5G. Τώρα, αντίκτυπο στα κέρδη. Δεν έχουμε σχετικές στατιστικές, αλλά βλέπουμε τα ωφέλη και για τους χρήστες, ε, τους επιχειρηματίες, αλλά και για τους απλούς πολίτες, εφόσον το κόστος της περιαγωγής έχει ε, εξαλειφθεί. Για το 5G είναι το θέμα της ευρείας ζώνης για όλους. Ε, εδώ Βεβαίως αυτό δεν υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σε ορισμένα μέρη υπάρχουν ε, δίκτυα ψηλή ταχύτητα με νευραίω δεδομένα, ενώ αλλού όχι. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει με τη δημογραφική κατάσταση τη κάθε χώρα. Στο Μπέρεκ και με τα NRA προσπαθούμε να, να, να βοηθήσουμε στη δημιουργία ε, ε, ε, επενδύσεων και κρατικών επενδύσεων εκεί όπου δεν υπάρχει κίνητρο για τις ιδιωτικές, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι κάθε πολίτης και εταιρεία στην Ευρώπη θα έχει πρόσβαση στην ε, μεγάλη ταχύτητα σε ευρεία ζώνη. Τέθηκε ερώτηση για το να μείνει κάποιο φάσμα για βιομηχανικούς σκοπούς. Κοιτάξτε, όταν έχουμε το φάσμα των 26 GHz, ε, το πώς αυτός ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί, αυτό το εξετάζουν οι NRA και οι διαχειριστές φάσματος. Η ιδέα είναι να χρησιμοποιηθεί χωρίς ε, χορήγηση άδειας ε, από συγκεκριμένους χρήστες. το θέμα της Γερμανίας που έχει βάλει κατά μέρος φάσμα για τις βιομηχανίες. Τώρα κατά πόσο αυτό είναι σωστό ή όχι εξαρτάται από την εθνική κατάσταση στη Γερμανία που έχουμε πολύ μεγάλους βιομηχανικούς χρήστες με μεγάλες εγκαταστάσεις που φτάνουν ε, στη, σε μέγεθος ε, πόλης κάποιες φορές. Εμείς στην Ιρλανδία από όπου προέρχομαι δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Δηλαδή το φάσμα που είναι διαθέσιμο για την Ήπεθρο ε, είναι πιο ενδιαφέρον για μας γιατί δεν έχουμε τέτοια μεγέθη. Ε, νομίζω πως η, βιομηχανία της κινητής τηλεφωνίας λέει αφήστε το σε εμά, εμείς θα δούμε πού χρειάζεται και πού όχι. Οι βιομηχανικοί χρήστες το χρειάζονται γιατί υπάρχουν κάποιες σημαντικές ε, ε, εφαρμογές. Ευχαριστώ. Να προσπαθήσω και εγώ να χρησιμοποιήσω σωστά το 1,5 λεπτό μου. Λοιπόν, κέρδη για τους ε, φορείς κινητής τηλεφωνίας. Ε, νομίζω πως ε, έχουν αντισταθμίσει καλά τα απώλειες από τα έσοδα της περιαγωγής. Τώρα για το κατά πόσο θα πρέπει να έχουμε ή όχι εθνικές αποφάσεις για το φάσμα 5G ε, για βιομηχανική χρήση δεν είναι μόνο η Γερμανία και η δική μου χώρα σκέφτεται να κάνει το ίδιο ε, και νομίζω ότι η άποψη ε, ανταγωνισμού είναι καλό το να έχουμε διαφορετικά είδη προμηθευτών στην αγορά να έχουμε συζήτηση με τους φορείς μας που λένε ότι ναι, δώστε μας τα όλα και εμείς θα φτιάξουμε σωστά την αγορά, έτσι λένε συνήθως. Αλλά το να υπάρχει μια άμεση παροχή είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο αξίζει τον κόπο να το χρησιμοποιήσουμε. Τώρα, για την κυβερνοασφάλεια, ε, αυτό που εμείς κάνουμε συνήθως για την ασφάλεια είναι ένας κανονισμός ακεραιότητας, κοιτάμε δηλαδή την ε, ασφαλή χρήση του δικτύου, την ασφαλή δυνατότητα ενημέρωσης του δικτύου, ενημέρωσης των κωδικών στο σύστημα, γιατί πολύ συχνά το πρόβλημα είναι ο χειρισμός συστημάτων όταν κάνεις την ενημέρωση. και επίσης να έχουμε καλά συστήματα για αξιόπιστες ε, αναφορές. Και μαθαίνουμε από αυτά καθημερινά. Μπορούμε να αναπτύξουμε αρχές κυβερνοασφάλειας σε αυτούς τους τομείς ε, που είναι πιο κοντά στις δικές μας αρμοδιότητες. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Γκάλφρη, κύριε Σερπλάμ, κύριε Ινέση. Είναι 11 και 4. Ε, τέλεια τα πήγαμε από άποψη χρόνου. Σε πολύ ενδιαφέροντα δε τα όσα μας είπατε και οι απαντήσεις που δώσατε στις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που ακούσαμε. Σας ευχαριστώ ε, πολύ και θα τα ξαναπούμε σύντομα. So next item, last item on the agenda. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης για ε, τώρα το ε, πρωί την ανταλλαγή απόψε με τον ε, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, κύριο Ζαμπιέ Μπουγνιού, και με τον καθηγητή Άντσιο ο οποίος είναι διευθυντής στο Ινστιτούτο Αλφρεντ Φίγνα εργάζεται για θέματα που αφορούν τις κλιματικές αλλαγές, την βιοχημία και τη βιοπικιλότητα στον Αρκτικό. Καθώς λοιπόν ετοιμαζόμαστε στη λήξη της δεύτερης θητείας σας, ε, καθώς προετοιμάζουμε την επόμενη χρηματοδότηση για το, για το ερευνητικό πρόγραμμα Horizon ε, Ευρώπη, θα θέλουμε να ακούσουμε ε, τις απόψεις σας σχετικά με το πώς μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε ε, το χρηματοδοτικό περιβάλλον ε, για την έρευνα και επίσης θα θέλαμε να ακούσουμε κύριε καθηγητά Μποίτσιους το πώς η χρηματοδότηση, το πώς η χρηματοδότηση από το Συμβούλιο Έρευνας βοήθησε την ε, έρευνά σας, ε, την καριέρα σας ε, και το πώς βοήθησε στο να βρεθούν λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Έχουμε συνολικά μία ώρα και 15 λεπτά για το θέμα αυτό, για τη συζήτηση αυτή και θα ήθελα να δώσω αρχικά το λόγο σε εσάς, καθηγητά ε, Μπουγινιού. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Το ευχαριστώ ε, τον ε, Αντιπρόεδρο κύριο Πέτσασεν τα αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Ήταν μεγάλη μου τιμή ε, που από τον Ιανουάριο του 2014 για έξι σχεδόν χρόνια ήμουν διευθυντή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνα την πρώτη φορά που ήρθα σε αυτή την ε, επιτροπή ε, συστήθηκα ε, σε εσά και παρουσίασα τις προτεραιότητες του Συμβουλίου. ερχόμουν τακτικά στο Κοινοβούλιο και πάντοτε έβρισκα υποστηρικτές εδώ. Το, έρευνα, το ενδιαφέρον σας για την έρευνα και ιδιαίτερα για το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο Έρευνας ήταν έντονο και πάρα πολύ συχνά οι παρεμβάσεις σας ήταν πολύ σημαντικές. Καθώς λοιπόν πλησιάζω στο τέλος της θητείας μου ως ε, πρόεδρος ε, του Συμβουλίου θα ήθελα και πάλι να σας ενημερώσω και να σας πω και να σας υπενθυμίσω για ποιο λόγο δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνα. Το 2007 ο πρώτος ε, πρόεδρος του Συμβουλίου έδωσε μία ομιλία υπό την καγκελαρία της κυρίας Μέρκελ, απέστειλε ένα μήνυμα το οποίο ήταν ευθυγραμμονισμένο με τους, ε, με τις προσπάθειες για τη δημιουργία του συμβουλίου. Ο Διευθυντής τότε είχε πει ότι το ε, σημαντικό πλεονέκτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για το μέλλον θα είναι να επενδύσουμε στην έρευνα που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της, ε, ε, του πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ο μόνος τρόπος για να διαβαλουσιούμε ότι οι επενδύσεις θα αποφέρουν θα είναι η αριστεία. Πολλά έχουν αλλάξει από το 2007, πολλά όχι προς το καλύτερο, όμως πιστεύω ότι αυτά τα λόγια είναι ακόμα πιο σημαντικά σήμερα. Σε σύγκριση με άλλε περιοχές του πλανήτη η Ευρώπη είναι πιο πλούσια, έχει καλύτερη ποιότητα ζωής και αυτό οφείλεται όχι στους αριθμούς τη και τους φυσικούς τη πόρους αλλά ε, λόγω της παράδοσης μας ε, που ε, φτάνει στην αναγέννηση οπότε και αναζητούσαμε απαντήσεις, να βρούμε λύσει και να τι χρησιμοποιήσουμε ώστε να διευκολυνθεί η ζωή των συμπολιτών μας έχουμε ε, την ικανότητα να διαχωρίσουμε την χρήσιμη από την άχρηστη ε, γνώση και έτσι λοιπόν θα πρέπει να υποστηρίξουμε την καινοτομία για το μέλλον. Η μακροπρόθεσμη ε, χρηματοδότηση για την έρευνα θα πρέπει να διατηρηθεί διότι αυτή ήταν η πηγή πολλών κοινοτομιών στο παρελθόν. Διότι διαφορετικά θα κινδυνεύσουν, θα θέσουμε σε κίνδυνο τους ε, σπόρους της ε, καινοτομία. Και αυτό το βλέπουμε, για παράδειγμα, με την έρευνα που κάνουμε στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή τη στιγμή οι κυβερνήσεις ε, αλλά και οι επενδυτές θέλουν να χρηματοδοτήσουν τον τομέα αυτόν και βασίστηκε στην δίψα που είχαμε για την προώθηση του τομέα αυτού. Την δεκαετία του 80 και 90 υπήρξε χρηματοδότηση ε, σχετικά με την τεχνητή, ε, ε, τεχνητή νοημοσύνη. Όμως στη συνέχεια μία σειρά ερευνητών συνεχίσαν, συνέχισαν τις έρευνες σε αυτόν τον τομέα και κατόρθωσαν να φέρουν σε νέο επίπεδο ε, την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή τη στιγμή, 30-40 χρόνια αργότερα, η τεχνολογία αυτή επηρεάζει την ε, κοινωνία. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε νέα όρια τώρα που αφορούν άλλε ε, διαστάσεις θα είναι σημαντικό λοιπόν η ε, πολιτική σχετικά με την έρευνα και την ε, καινοτομία να αναπτύξει αποστολέ ε, σε αυτόν τον τομέα. Όμω οι προκλήσει που έχουμε να αντιμετωπίσουμε παγκοσμίω είναι τεράστιε και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρξουν προσπάθειε από του ερευνητέ ούτω ώστε να κατανοήσουμε το τι συμβαίνει για πολύ καιρό υποτιμούσαμε τις αλλαγές που ε, θα υπήρξαν λόγω της ε, αντίληψης των βασικών των φαινομένων, ε, λόγω των κλιματικών αλλαγών και της σειράς ερευνών που έχουν γίνει γνωρίζουμε ότι το business as usual δεν πρόκειται να μας βοηθήσει. Έτσι λοιπόν δεν θα είχε λογική το να αφαιρέσουμε τη δυνατότητα στους Ευρωπαίους για αυτές τις σημαντικές έρευνες ε, θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο για τα επιστημονικά ε, μυαλά, ούτως ώστε να κάνουν ε, την, το σημαντικό τους έργο που πάντοτε μας εκπλήσει. Αυτό μπορεί να προέλθει, να προκύψει μονάχα από έρευνα εχμής. Και όλο αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα, μια δυνατότητα που θα τοποθετήσει την Ευρώπη στην κορυφή της ερευνάς εχμής. Αναφέρθηκε αυτό ήδη σε μια έκθεση του 2017 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας αναγνωρίζεται ως ένας παγκόσμιος παίκτη στον τομέα της επιστημονικής αριστείας χάρη στις δομές που έχουν ε, τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν παίξει ένα σημαντικό ρόλο ε, στην, ε, έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της αριστείας και της έρευνας στην επιστημονική κοινωνία. Ε, κοινότητα. Ταυτόχρονα έχουμε δει ότι οι νέοι ερευνητές της Ευρώπης έχουν ε, λάβει τη δυνατότητα να ε, καθορίσουν τους δρόμους που θα ακολουθήσουν χωρίς να τους επιβάλλονται επιλογές. Έχουν δοθεί έχουν ε, δοθεί επιχορηγήσεις σε 80 διαφορετικά ερευνητικά Ινστιτούτα. Πολλοί έχουν ε, ξεκινήσει έρευνες ε, για πρώτη φορά στην ακαδημαϊκή τους καριέρα και γι' αυτό το λόγο πολλοί εξ αυτών λένε ότι το Συμβούλιο έχει αλλάξει τη ζωή μου. Ε, περιλαμβάνονται 70.000 ε, μέλη στην έρευνα ΕΦΤΕ, στις ε, διάφορες έρευνες. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι τα αποτελέσματα έχουν ε, σημαντικές ε, συνέπειες όπως έχει ε, φανεί από την εκ των υστέρων αξιολόγηση δημοσιοποιήσεις από έρευνες που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Συμβούλιο έχουν 7 φορές μεγαλύτερες πιθανότητες να αναφερθούν σε άλλες έρευνες στη συνέχεια. Ορισμένα παραδείγματα ε, είναι ότι έχουν ε, κατορθώσει να κάνουν καινοτομίε ε, στον τομέα των ηλιακών συλλεκτών σε τομείς όπως αφορούν τις κοινοτόμες ουσίες, έχουν δημιουργήσει μοντάλα συστημικών κινδύνων στον χρηματοπιστωτικό τομέα και έχουν εξετάσει το πώς το κλίμα επηρεάζει την μετανάστευση η ανάγνωση των ανθρωπίνων συναισθημάτων από, ε, μηχανή, από μηχανές, οι έρευνα όσον αφορά τις ε, οπές. Επίσης, ε, υπήρξαν έρευνες σχετικά με το πώς ε, τα κύτταρα ε, απορροφούν το οξυγόνα, κάτι το οποίο μπορεί να αποτελέσει βάση για την αντιμετώπιση πολλών ασθενειών. Όλα αυτά είναι μερικά από τα όσα ε, ερευνητικά προγράμματα έχει χρηματοδοτήσει το Συμβούλιο Έρευνας. Η μακροπρόθεσμη συνέπεια λοιπόν του Συμβούλιο είναι ξεκάθαρη και έχουμε βοηθήσει και σε ε, βραχυπρόθεσμο επίπεδο. Ε, το Συμβούλιο εισήγαγε ένα πλαίσιο χρηματοδότηση το 2011 το οποίο δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει μια μεγαλύτερη προσέγγιση στις αγορές. Ε, έχουν δοθεί πάνω από χίλιες τέτοιες επιχορηγήσεις, έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές νέες εταιρείε χάρη σε αυτή τη χρηματοδότηση. Από πλευράς μου λοιπόν, λοιπόν χαίρομαι που μου δόθηκε η δυνατότητα να ε, βοηθήσω σε αυτήν τη σημαντική ε, επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2014 προτεραιότητά μου ήταν να διατηρήσω την ε, το υψηλό επίπεδο της ε, διαδικασίας επιλογής του Συμβουλίου Έρευνας, το οποίο δεν είναι μια απλή διαδικασία που θα πρέπει να λάβουμε δεδομένα. Λαμβάνουμε ετησίως 10.000 αιτήσει. Ε, χρειάζεται πολλούς χρόνους αξιολόγηση αυτών των, αυτών των αιτήσεων. υπάρχει μεγάλη ε, ζήτηση για ε, τους ε, ανθρώπους οι οποίοι αξιολογούν αυτές τις αιτήσει και θα πρέπει λοιπόν να τους αφιερώσουμε τον χρόνο μας. Όταν ξεκίνησε η θητεία μου, η θητεία μου το 2014 υπάρχουν τρει που θεωρούσα ότι θα μπορούσε να υπάρξει βελτίωση. Για παράδειγμα, η, η ισορροπία όσον αφορά την εκπροσώπηση των ε, φύλων. Ε, υπήρξε, ε, υπήρξαν, υπήρχαν πολύ λιγότερε αιτήσει από γυναίκε, όμω, χάρη στο σχέδιο περί τη ισότητα των φύλων θα ήθελα να σα αναφέρω ότι για την περίοδο 14-19 ε, το ε, ποσοστό επιτυχία είναι ίσο μεταξύ ανδρών και γυναικών. Επίση, εργαστήκαμε σκληρά ούτως ώστε να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των ερευνητών από τις ε, περιοχές της Ευρώπης που συμμετέχουν λιγότερο στην έρευνα τα τελευταία χρόνια το ε, Συμβούλιο Έρευνας έχει ε, δημιουργήσει την, ε, τη χρηματοδότηση για τους επισκεπτόμενους ερευνητές. Έχω επισκεφθεί όλες τις χώρες κράτη-μέλη εκτός από μία και έχω πάει, ε, θα πάω στην Ουγγαρία, στην ε, Σλοβενία, Σλοβενία τις επόμενες εβδομάδες ε, και τα ποσοστά συμμετοχής έχουν, παρακολουθούνται καθόλου την διαδικασία αξιολόγησης. Γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να κάνουμε πολλά ακόμα, όμως από το 2014 οι έρευνες σε Τσεχία, Ελλάδα, Σλοβεκία έχουν δει μια αύξηση πάνω από το μέσο όρο και από το 2014 η έρευνα σε Ρουμανία, Λιθουανία, Σερβία, έχουν λάβει χρηματοδότηση για πρώτη φορά. Ε, και επίσης ανακοίνωσα ε, τις, τα, ε, τις αιτήσει για έρευνα και ε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε συνεργασία με ε, ερευνητικά Ινστιτούτα, ε, με ερευνητικά Ινστιτούτα σε όλο τον πλανήτη. Όλες αυτές οι δράσεις σε διάφορα πεδία δείχνουν το πόσο σημαντικό είναι να κρατήσουμε αυτό το θετικό momentum και θα πρέπει συνεχώς να αξιολογούμε τις δράσεις μας με πλήρη διαφάνεια και όποτε είναι αναγκαίο να προσαρμοζόμαστε. Παρ' όλα αυτά όμως μεταγιώνω για ένα πράγμα ως έχαμε ε, πολλές προτάσεις τις οποίες όμως δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε. Από την έναρξη του ε, Horizon 2020 από το 2014 ε, πολλά ε, προγράμματα έχουν ε, θεωρηθεί άριστα από το πάνελ μας παρόλα αυτά όμως δεν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν. Αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο μπορεί να χρηματοδοτήσει το 12% των προτάσεων που λαμβάνουμε. Αν μπορέσουμε να φτάσουμε το 15% τότε θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις μη χρηματοδοτούμενες ε, προτάσει ε, που θεωρούμε πάρα πολύ καλέ αυτέ είναι οι προτάσει του Συμβουλίου Έρευνα. Κλείνοντα, θα ήθελα και πάλι να σα ευχαριστήσω για τι ε, δυνατότητες που μου δώσατε να σας παρουσιάσω το που βρισκόμαστε. Ο ε, διαδοχός μας, θα, ο διαδοχός μου θα αναλάβει το ε, Ιανουάριο του 2020. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ρώμη. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι θα πρέπει να αποφασιστεί ο προπολογισμό για το Horizon 2020. Σίγουρα θα είναι ένας δύσκολο αγώνας που έχει ήδη ξεκινήσει και ελπίζουμε ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Το Κοινοβούλιο έχει δηλώσει ότι θα υποστηρίξει ε, ένα προϋπολογισμό 20 ε, δισεκατομμυρίων ε, και θα πρέπει να επιτύχουμε τους στόχους μας ε, δεν θα πρέπει να έχουμε μέτριες φιλοδοξίες, θα συνεχίσουμε αυτό τον αγώνα ε, για τους ε, Ευρωπαίους ερευνητές και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τα παράτητα μέσα για ένα βιώσιμο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπουργινιόν και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο σε εσάς κυρία Άντζε Ποέτσιους ναι, μπορώ και εγώ να δείξω τις διαφάνειές μου. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να παρουσιάσω το παράδειγμα της δικής μου καριέρας στον τομέα της έρευνας για να διευκρινίσω ε, τα ζητήματα αυτά. Η αποστολή μου λοιπόν είναι το, το κλίμα στην Ακτική. Έχω λάβει και ένα βραβείο σχετικό. Ε, έψαχνα να βρω ποιο είναι το πιο καταλημμένο βακτήριο στους ωκεανούς. Ε, μπορεί να, να, θέλει, να θέλει να το ξέρει κανείς ή να θέλει να μάθει γιατί δεν το ξέρει κανείς. Θέλω να κάνω τη διαφορά διότι το περιβάλλον μας το, το διαχειρίζονται, ε, είναι μάλλον γεμάτο μικρόβια. Έχουμε όμως τόσους ωκεανούς, ε, τόσες εκτάσεις και δεν ξέρουμε ποια μικρόβια υπάρχουν εκεί. Ήμουν εκεί λοιπόν ε, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2012 είχα την ευκαιρία να μελετήσω έναν τομέα σε μια περιοχή όπου κανείς δεν είχε ε, μελετήσει στα βάθη της θάλασσας τα μικρόβια είχα την ευκαιρία να δω πράγματα που δεν είχε δει κανείς. Ε, μπορούσα να δω ποια βακτήρια είναι σημαντικά στον κύκλο ζωής ε, και βεβαίως ε, επικεντρώθηκα στα θέματα τη γενικότερα. Δεν θα μιλήσω τώρα βεβαίως για το παρελθόν και το τι έκανα, διότι έχει τελειώσει εκείνη η έρευνα. Θα ήθελα όμως να πάω να κοιτάξω προς το μέλλον και να σας πω πώς συνδέεται η αριστερή ε, και η περιέργεια του ανθρώπου με τις αποστολές αυτές. Υπάρχει μια αποστολή αυτή τη στιγμή που λέγεται Μοσαϊκ και εδώ βλέπετε ότι στην αρχή του έτους αυτή η αποστολή θεωρήθηκε ίσως η πιο το πιο σημαντικό βήμα στη διεθνή επιστήμη για το όλο έτος. Τι ακριβώς, ε, περί πρόκειται. Σας παρακαλώ να καθίσετε να σκεφτείτε κι εσείς λίγο την περιοχή του, βο, Βόρειου Πόλου, ε, το θέμα της ε, ε, συνδεσιμότητας της Ευρώπης με το Βόρειο Πόλο. Γνωρίζουμε για τον καιρό, γνωρίζουμε για το κλίμα, αλλά είναι και μια μελλοντική, μελλοντική περιοχή για απασχόληση, για μεταφορές, επειδή αλλάζει το κλίμα. Αυτή τη στιγμή ε, έχουμε υποστήριξη και από ε, άλλες, ε, άλλους ερευνητές. Ε, για πρώτη φορά προσπαθούμε να βρούμε πώς λειτουργεί ο χειμώνα στην Αττική, πώς αλλάζει το κλίμα, πώς θα, αλλάξει το καλοκαίρι. Ε, τέτοιου είδους ερωτηματικά δεν έχουν τεθεί, τέτοια είδους έρευνα δεν έχει λάβει χώρα με τις σύγχρονες υποδομές, τη σύγχρονη τεχνολογία. Εδώ βλέπετε ερευνητές σε διάφορους τομείς που χρησιμοποιούν τα εργαλεία τους έτσι ώστε να μπορέσουν να γίνεται και ολόκληρο έτος. για να μετρήσουν τα πάντα. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε αυτό το τεράστιο, την τεράστια πρόκληση, έτσι ώστε να μπορέσουν όλοι να επιστρέψουν οι άνθρωποι αυτοί ζωντανοί. Ένα ε, δίκτυο ερευνητών θα δώσει στοιχεία για τις επόμενες γενιές ε, που είναι απαραίτητα για να καταλάβουμε το ρόλο ε, του Βορείου Πόλου και της Ακτικής γενικότερα για το Βόρειο Εμισφαίριο. Χαίρομαι και είμαι περήφανη που το Ινστιτούτο μου και οι άνθρωποι από παντού ε, κάνουν αυτήν τη μεγαλύτερη αποστολή που υπήρξε ποτέ για το πιο κρίσιμο ζήτημα της εποχής μας. Πώς οι ωκεανοί και οι πολικές περιοχές καθορίζουν το κλίμα στον πλανήτη Γη. Ξεκίνησε το 12 Σεπτεμβρίου αυτή η αποστολή και το πλοίο αυτή τη στιγμή έχει παγώσει, είναι σταματημένο στον πάγο, προχωράει αργά ε, και θα μπορέσει να φτάσει ως το Βόρειο Πόλο. Αυτός είναι ο στόχος και εκεί όπου υπάρχει ε, πάγος σκληρός θα υπάρξουν διάφορα στρατόπεδα, άλλα πλοία θα αλλάξουν ε, πληροφορίες οι επιστήμονες. 600 άτομα θα συμμετάσχουν σε αυτή τη μεγάλη εμπειρία και μπορούν να θέσουν ερωτήματα ε, σχετικά με την έρευνα αυτή, τι σημαίνει η τι σημαίνει για τη ζωή μας, ε, η χημεία στην ακτική η ατμόσφαιρα και βεβαίως ποιες είναι, ποια είναι η μετρολογική ε, αλληλουχία. Δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό, αυτή η αποστολή αν δεν ήταν πολλά ευρωπαϊκά δίκτυα και πολλές χώρες ε, με τους παγοθράφτες τους, τα παγοθραφτικά τους, υπάρχει ένα δίκτυο παγωτραυστικών και ένα σχετικό πρόγραμμα που μας επιτρέπει γρήγορα να βρούμε την μηχανική υποστήριξη όταν κάνουμε τέτοιου είδου έρευνε. Το που βλέπετε εδώ είναι ε, το, ο πυρήνα αυτού του κέντρου αριστεία για τέτοιου είδου αποστολέ στου ωκεανού και στι πολικέ περιοχέ, για τα οποία λίγα πράγματα γνωρίζουμε, αλλά είναι πολύ σημαντικά για το μέλλον μα. Βλέπετε εδώ νέου ανθρώπου, επιστήμονε που προέρχονται από την Ευρώπη, από αλλού, μπορεί να χρησιμοποιήσουν τι σχολέ του, τις υποτροφίες τους, κάνουν PhD, κάνουν μια καριέρα. Ε, αλλά αυτή, την αποστολή, αυτή η αποστολή θα μιλάμε για αυτήν για πάντα, διότι τα στοιχεία που θα προκύψουν με αυτόν τον τρόπο ε, θα ανοίξει την πρόσβαση σε δεδομένα που θα αλλάξουν τη ζωή μας. Αυτό το γνωρίζουν ε, και εγώ με μεγάλη χαρά συζήτησα μαζί τους όταν ξεκίνησε η αποστολή το Σεπτέμβριο του 2019 πριν από δύο μήνες περίπου. Εκεί βρίσκεται αυτή τη στιγμή το πλοίο και μπορείτε να δείτε τα πρόσωπα χαρούμενων επιστημόνων. Δεν βλέπετε βέβαια πόσο χαρούμενοι είσαστε, διότι είναι, διότι είναι παγωμένοι. Αλλά υπάρχει αυτή η εικόνα της ευρωπαϊκής αριστείας και της διεθνούς συνεργασίας. Ε, μπορεί να ερχόμαστε από παντού στην Ευρώπη, αλλά εκεί, στον πολιτικό χειμώνα, ε, τα, ε, ε, όλοι παγωμένοι θα είμαστε και το ίδιο θα μοιάζουμε. Θα συμμετέχουμε σε μια ίδια αποστολή έρευνα. Διότι η περιοχή τη ακτική είναι ένα νέο τομέα, ένα νέο πεδίο που πάει πέρα πια από την περιέργεια. Είναι μια από αυτέ τι περιφέρειε που από γεωπολιτική πλευρά ε, γίνονται μεγάλε ζητήσει για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση για να αλλάξει ε, η ζωή των ανθρώπων που ζουν εκεί. Τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι ζουν εκεί. Δεν είναι έρημο. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα για, για τον Αρκτικό ωκεανό και αυτήν την ε, λεκάνη που θα ε, μελετήσουμε τα, επόμενα χρόνια. Θα μοιραστούμε τις ιστορίες των ερευνητών, θα υπάρξει πρόσβαση στην επιστημονική μέθοδο με ένα blog καθημερινό, ε, υπάρχει, υπάρχει επικοινωνία ε, μεταξύ επιστημονών, ε, υπάρχουν εκεί μέσα ενημέρωσης, θα κυματογραφηθούν όλα αυτά και θα έχουμε ντοκουμέντα στη συνέχεια. Ε, τα οποία θα είναι χρήσιμα και τι επόμενε δεκαετίες. Θα ήθελα να σας πω ότι τέτοιου είδους ε, χρήση τη επιστημονική έρευνα για να σπάσουμε τα σύνορα τη γνώση, ε, που καθορί, γνώσεις που καθορίζουν το μέλλον μας, αυτά είναι στο DNA μας. Μπορεί να μην το γνωρίζετε, αλλά βρήκα στοιχεία ε, ότι έχει, έχει γίνει έρευνα σε πολλές χώρες της Ευρώπης για, για τον Μπόριο Πόλο. Κάποτε όλοι ήθελαν να πάνε εκεί όλοι ήθελαν να καταλάβουν τι συμβαίνει στο Βόρειο Πόλο, τι κρύβει ο Βορειο Πόλος ε, για μας ε, σε επίπεδο πόρων. Το είχε κάνει αυτό ο Φρίτχοφ Νάνσεν τότε, το 19ο αιώνα. Ε, είπε, οι επιστήμονες πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε, διότι σε 100 χρόνια δεν θέλει ο κόσμο να ξέρει πόσο κρύο, η πόσο κρύα ήταν η αποστολή μας. ήταν βεβαίω οραματιστή αυτός, ε, διότι όλοι τώρα κοιτάζουμε όλα αυτά τα όργανα για να δούμε πόσο γρήγορα και γιατί τόσο γρήγορα ζεσταίνεται ο ωκεανός ε, και η αρκτική περιοχή ε, δύο-τρεις φορές πιο γρήγορα από στον υπόλοιπο κόσμο. Μέρος αυτής της περιέργειας που οδήγησε σε αυτήν την επιστήμη και που κάνουμε χάρη στην αριστεία μας έχει να κάνει με την, το, το ζήτημα ενός βιώσιμου πλανήτη και του μέλλοντος της ζωής μας. Ως Ευρωπαίοι επιστήμονες παρουσιάζουμε αυτές τις γνώσεις σε όλους όλους όσους ε, έχουν θέσεις ισχύω. Ε, σημειώνεται πρώτος, πιστεύουμε ότι η Ευρώπη ε, θα πρέπει να συμφωνήσει για ένα μορατόριο στην ε, να προστατεύσουμε κάποια είδη εκεί. Από την άλλη υπάρχουν ε, απειλές ε, όπου δεν ξέρουμε πώς θα τον αντιμετωπίσουμε όπως ε, το permafrost, ε, όπου το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι σε διεθνές επίπεδο να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε ε, το, τα ενεργειακά μας συστήματα, η μόλυνση, τα πλαστικά, όλα αυτά λαμβάνουν χώρα σε μια περιοχή για την οποία γνωρίζουμε λίγα πράγματα και όπου οι επιστήμονες φτάνουν στο συμπέρασμα ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν ε, όσο, προχωρήσουμε όσο γρήγορα όσο αλλάζουν τα πράγματα. Θα τελειώσω με δυο τρει ακόμα διαφάνειας για να σας πω τι παρατηρούμε ε, αυτή τη στιγμή βελτιώνουμε το μελλοντικό μοντέλο για να καταλάβουμε πώς τα πολιτικά συστήματα αλλάζουν το κλίμα μας. Ε, πάμε πίσω στο παρελθόν και εδώ βλέπετε άλλη μια φανταστική αποστολή στην πολική περιοχή, το οποίο χρηματοδοτείται από αυτό το πρόγραμμα και από το επόμενο. Ε, είναι το πιο, το πιο, το πιο παλιό παγετώνες της ε, για να δούμε τι γίνεται με τη διακύμανση του διεξιού του άνθρακα. Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή 400, κάτω από 400, 400 ppm και βλέπετε τι είχε γίνει πριν τη βιομηχανοποίηση. Ε, ε, με την ανθρώπινη εξέλιξη ποτέ δεν είχαμε φτάσει σε τέτοια συγκέντρωση διευσίου του άνθρακα όπως σήμερα. Αν πάμε πίσω στο χρόνο, εάν και αν προβλέψουμε το μέλλον μας και βλέπετε εδώ την κίτρινη γραμμή σε ό,τι αφορά την ε, θερμοκρασία που έχει να κάνει με την ανθρώπινη εξέλιξη, βλέπετε ότι στο μέλλον με ανάλογα με τον δρόμο που θα ακολουθήσουμε, βλέπετε τι θα γίνει η θερμοκρασία. Και βλέπετε τι έχει γίνει στο παρελθόν. Κάποτε είχαμε 400 ε, ppm ο τότε όμω ήταν 20 μέτρα πιο πάνω η θάλασσα. Ήταν πολύ μικρότερη κάλυψη από παγετών, ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή την οδό ακολουθούμε και πρέπει να πάρθουν αποφάσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτή η μικρή λοιπόν αποστολή, αυτό το ταξίδι ε, στην έρευνα αυτή ε, θέλω να δώσει κάποια κίνητρα προς εσάς για να σκεφτείτε πώς θα οικοδομήσουμε το μέλλον μας ε, υποστηρίζοντας την έρευνα ε, όντας ενωμένη ε, στα πλαίσια της έρευνας. Εδώ βλέπετε ένα γράφημα που, που δείχνει και πάλι την πρόοδο την, την της και το τι πρέπει να γίνει. Η επιστήμη είναι αυτή που θα δείξει τον δρόμο. Ε, είναι απαραίτητο να σκεφτούμε ότι η επιστήμη είναι μέρος του μέλλοντος της Ευρώπης. Και ε, αυτά σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και ελπίζω ε, να σας αρέσει αυτή η εικόνα του πόλα Στέρν που είναι εκεί σταματημένο στον πάγο ε, με πολλούς ε, συνάδελφους Ευρωπαίους εκεί. Uh, uh, σας ευχαριστώ και τώρα θα ακούσουμε ερωτήσεις των συντονιστών και προς τους δυο σας. Η κυρία Καρβάλιο πρώτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ καθηγητά Μπουργινιό που είστε εδώ και για όλη σας την δουλειά στο ERC. Θεωρούμε ότι το ERC και το Erasmus είναι μάλλον τα πιο επιτυχή ευρωπαϊκά προγράμματα όπως ακούμε από τον κόσμο στη διάρκεια των ε, ε, προεκλογικών μας εκστρατιών. Είχατε εξαιρετικά αποτελέσματα όσον αφορά τις δημοσιεύσεις ε, και τις εφαρμογές αυτών των γνώσεων. Είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να είμαστε περήφανοι. Τώρα, ωστόσο, ξεκινάμε τα τελικά στάδια του το Horizon Europe και πρέπει να εξετάσουμε ποια σημεία μπορούμε να βελτιώσουμε. Και θα ήθελα να ρωτήσω τη γνώμη σας για δύο πράγματα. Πρώτον, τα αποτελέσματα του ERC θα μπορούσαν να εσωματωθούν καλύτερα στις άλλες, στα άλλα κομμάτια του Horizon. Δηλαδή, οι αποστολές ε, στο μέλλον, το EIT, Βλέπω πολύ συχνά πως ε, εσείς ε, έχετε project σε άλλα κομμάτια του Horizon 2020 που δεν χρησιμοποιούν τα μοντέλα Δηλαδή δεν υπάρχει ένας αγωγός, είναι κάτι για το οποίο αγωνιζόμαστε ε, εδώ και χρόνια να δημιουργηθούν δηλαδή ε, οριζόντια αγωγή ανάμεσα στα προγράμματα πλαίσια ώστε να διαδίδονται τα, τα πορίσματα. Πάντως το ERC είναι ένας πολύ σημαντικός τρόπος, καλός τρόπος για να ε, προχωρήσουμε και στα άλλα τμήματα γιατί έτσι γίνονται φανταστικές έρευνες και ε, συχνά υπάρχουν ε, πολλές εφαρμογές. χωρίς να έχουμε πάντοτε όμως την επιστημονική βάση που μπορεί να υπάρχει για την ε, έρευνα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεύτερο ερώτημα αφορά το ποσοστό επιτυχίας. Είπατε πως υπάρχει ένα ποσοστό ε, επιτυχίας και αριστείας για τις προτάσεις που είναι καλές για να χρηματοδοτηθούν, αλλά δεν έχουμε αρκετά χρήματα. Για να είμαστε ρεαλιστές, όπως ξέρετε εδώ έχουμε ένα αίτημα για να αυξήσουμε τον προπολογισμό και κάνουμε ό,τι μπορούμε γι' αυτό. Αλλά ακόμα και στα καλύτερα, με τα καλύτερα σενάρια, η αύξηση του Horizon Europe θα είναι δεν θα είναι αρκετοί ώστε να χρηματοδοτηθούν όλες οι εξαιρετικές προτάσεις που εσείς αξιολογείτε εγώ πολλά χρόνια υπερασπίζομαι και έχω μάλιστα συντάξει και σχετική έκθεση ενώ ήμουν ε, ακόμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια έκθεση όπου πρότεινα και, α, και νομίζω πως έχετε ξεκινήσει να το κάνετε αυτό, να συνεργαστείτε λοιπόν με άλλους χρηματοδότες. Νομίζω πως ήδη το κάνετε αυτό, δηλαδή κράτη-μέλη, ε, με δημόσια χρήματα, περιφερειακά κονδύλια, ιδιωτικά ιδρύματα, ώστε με βάση συγκεκριμένα πρωτόκολλα να μπορούν να χρηματοδοτήσουν ε, κάποιο ε, κομμάτι αυτής της εξαιρετικής εργασίας. Γιατί όλα ε, η προετοιμασία για κάθε πρόταση είναι μεγάλη προσπάθεια. Πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση και εκεί είναι μεγάλη η προσπάθεια. Θα μπορούσε αυτός λοιπόν να είναι ένας τρόπος να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε περισσότερο τους ε, εξαιρετικούς μας ερευνητές μέσω της συσχέτισης μεταξύ άλλων ε, χρηματοδοτών και του ERC. Θα ήταν άλλο ένα πλεονέκτημα λοιπόν, ναι, ολοκληρώνω, ώστε να δημιουργηθεί ο ευρωπαϊκός χώρος έρευνας. Όλοι μαζί να συνεργαστείτε ώστε να χρηματοδοτείτε την καλύτερη δυνατή έρευνα δημόσιος και ιδιωτικό τομέα. Εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία στις προσπάθειές σας και εμεί σας ευχαριστούμε. Ο κύριος από το Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Μπουρκίνιο και να τον ευχαριστήσω για τη δουλειά που κάνει. Έχει αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις και με χαρά τον είδαμε και στη Ρουμανία και θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΕΣΥ για τη βοήθεια που μου προσέφερε στην προετοιμασία της έκθεσης στο Horizon 2000. Ξέρω πως υπήρχαν, υπήρξαν προκλήσεις, συζητήσεις, πολλά πράγματα που μάλλον θα μπορούσαν να, να έχουν γίνει καλύτερα, αλλά ελπίζουμε ότι τα πράγματα που διορθώσαμε στο Horizon Ευρώπη θα ε, τεθούν σε εφαρμογή γιατί έτσι θα υπάρχει μεγαλύτερο φάσμα για την εφαρμογή των κανόνων για τη χρηματοδότηση. Έχουμε τα κριτήρια ε, αριστείας επίσης που πιστεύω πως είναι τα καλύτερα, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα ότι δηλαδή έχουμε λιγότερα χρήματα στη διάθεσή μας και θα πρέπει να περάσουμε από τις διαπραγματεύσεις του για το PDP και θα δούμε πόσα χρήματα θα μείνουν τότε και επί τη βάση αυτών των ποσών θα πρέπει να σκεφτούμε στο επίπεδο του ERC με τον νέο πρόεδρο για το πώς ακριβώς θα γίνουν στη συνέχεια τα πράγματα. Πώς δηλαδή θα μπουν στην άκρη τα διαθέσιμα κονδύλια. Υπάρχουν πολλές φιλοδοξίες, θέλουμε να χρηματοδοτηθούν πολλά projects, αλλά πρέπει να δούμε και μειώσει σε πολλά άλλα project. Περικοπές γιατί ε, μπορεί κάποια κράτη να μην μπορούν να ωφεληθούν από τα χρήματα αυτά. Αν και είναι σημαντικό να δούμε projects από ολόκληρο τον κόσμο, είναι σημαντικό τώρα να δούμε πώς θα βρούμε τα χρήματα που χρειαζόμαστε. Ενώ ταυτόχρονα Υπάρχουν ε, επιτυχείς ε, περιπτώσεις που δεν ακούγονται όμως αρκετά, γιατί έχουν υπάρξει αυξήσεις στις δαπάνες, Όμως δυστυχώς η πτυχή των δημοσίων σχέσεων δεν έχει αναπτυχθεί αρκετά ώστε να διαδίδονται αυτές οι επιτυχίες. Οι επενδύσεις λοιπόν στη βελτίωση της ζωής των Ευρωπαίων πολιτών μέσω της έρευνας είναι κάτι το εξαιρετικά θετικό. Γι' αυτό και λυπάμαι που υπάρχει διαφορά, μεγάλη διαφορά, μάλιστα ανάμεσα στην έλλειψη των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα για το οποίο θα πρέπει να συνεχίσουμε να μιλάμε, γιατί ξέρω ότι μια από τις δικές σας επιθυμίες και επιθυμία του ERC, και θα πρέπει να δούμε τι λέει ο νέος πρόεδρος γι' αυτό, είναι ακριβώς ότι η αριστεία είναι το κριτήριο κλειδί η αριστεία οπουδήποτε και αν βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρηματοδοτείται καταλήλω. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω ακόμα μια φορά κύριε καθηγητά για όλα όσα κάνατε. Thank you so much, Mr. Nika. Now from Ευχαριστούμε πολύ. Από το Renew η κυρία Χλαμπάγιοβα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Όταν μιλάμε με ερευνητές παγκοσμίου επίπεδου, πάντοτε αναγνωρίζουν τη σημασία της χρηματοδότησης ε, ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν είναι μια ευρωπαϊκή επιτυχία. Εμένα μου αρέσει πολύ ο τρόπος που έχει διαστηθεί αυτός ο οργανισμός ως έναν εξάρτητο επιστημονικό συμβούλιο με δική σας στρατηγική, δικό σας πρόγραμμα εργασίας, δική σας επικοινωνία. Όταν όμως συζητάμε την έρευνα και την ανάπτυξη στην Ευρώπη και την καινοτομία στην Ευρώπη, ξεχνάμε πως η χρηματοδότηση της καινοτομίας είναι ένα μικρό κομμάτι της γενικής χρηματοδότησης για την έρευνα και την καινοτομία στην Ευρώπη. Το ορίζον Ευρώπη μάλλον θα είναι μόνο το 8 με 10% του συνολικού των δημόσιων δαπανών ε, για την έρευνα και την καινοτομία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άρα λοιπόν ε, θα πρέπει να δούμε και ποιο είναι το επίπεδο δωρεών. Άρα λοιπόν το ερώτημά μου είναι τι κάνει η ε, το οργανισμό σας για να γνωστοποιήσει τα πορίσματα και στα εθνικά κράτη, να κινητοποιήσει τα κράτη-μέλη ώστε να χρησιμοποιήσουν και να έρθουν πιο κοντά στο, και, στον στόχο του, του ΑΕΠ. Έπειτα, έχουμε πολλές αποστολές. Αυτό ήταν στο παρελθόν. Το Συμβούλιο πώς θα μπορέσει να συμβάλλει. Και εσείς, γιατί πραγματικά θαυμάζω την εργασία σας, δεν θα μπορούσα να κάνω αυτή τη δουλειά εγώ, μόνο παρακολουθώ τις δικές σας παρουσιάσεις. Αν όμως είχατε μια ευκαιρία να αλλάξετε ένα πράγμα όσον αφορά τις επιχορηγήσεις για τους ερευνητές, τι θα αλλάζατε. Ευχαριστώ Ματίνα. Από τους πράσινους η κυρία Ντάουριν. Τώρα, ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ και τους δύο που ήρθατε σήμερα και για τις ενδιαφέρουσες σας εισηγήσει. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την ε, κυρία Μπότης. πραγματικά φοβερή εμπειρία που είχατε ως ερευνήτρια και οι πληροφορίες που μας δίνετε μας κάνουν ε, να ταρακουνηθούμε σε σχέση με την έρευνα για το κλίμα και Γι' αυτό και θα θέσω ερώτηση στον κύριο Μπουργκινιό. Ως πράσινοι, εμείς θέλουμε πολύ να εξασφαλίσουμε πως θα επιτύχουμε το 35% για το οποίο έχουμε τώρα δεσμευθεί το 35% της ε, έρευνας το ορίζον ε, Ευρώπη. Το 35% λοιπόν να πάει σε θέματα έρευνας κλίματος. Ξέρω πως ο οργανισμός σας είναι ανεξάρτητος και ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το, τη δυνατότητα προγραμματισμού του προϋπολογισμού για να πιέσουμε για αυτό το 35%. Πιστεύω όμως που το CRC θα πρέπει να παίξει εκεί σημαντικό ρόλο. Και μια, ένα από τα επιτεύγματά σας, για παράδειγμα, είναι το να έχετε αυτήν την ισότητα ε, των φύλων και θέλω να ρωτήσω πώς θα αντιμετωπίσετε στο μέλλον το θέμα των κλιματικών δαπανών και πώς αυτό θα ε, μπει μέσα σε όλες τις πολιτικές του ERC. Έχετε πρόταση λοιπόν για συγκεκριμένα μέτρα τα οποία μπορεί να εφαρμόσει το ERC ώστε να συμβάλλει στην έρευνα για τις κλιματικές δαπάνες πάνω από τα κριτήρια επιλογής δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Τσονόφσκι από το ECR και έτσι θα κλείσουμε το γύρο των συντονιστών και μετά έχουμε και διάφορους άλλους συναδέλφους που θέλουν να θέσουν ερωτήσεις. Ο κύριος Στοζανόφσκι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μπουργκινιόν για τις εξαιρετικές του δραστηριότητες σε βάθος χρόνου ε, ξέρω πως ε, έχει να κάνει ένα γύρο των κρατών μελών και των νέων των μελών. Πώς λοιπόν μπορεί να αξιολογήσει την αύξηση των δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η δική μας Επιτροπή ΙΤΡΕ συχνά και τακτικά έχει θέσει ερωτήσεις ε, και έχει απασχοληθεί με το θέμα της ανισότητας για το πώς ορισμένες χώρες καταφέρνουν να χρησιμοποιήσουν και να απορροφήσουν τα κονδύλια του Horizon. Ιδιαίτερα τα νέα κρατημέλη δεν τα καταφέρνουν τόσο καλά. Και αυτό όχι γιατί δεν έχουν το κατάλληλο προσωπικό, μπορεί να υπάρχουν ιστορικοί λόγοι στο οποίο να οφείλεται αυτό. Ε, ακούω Οπότε ε, θέλω να θέσω την εξή ερώτηση. Ποια είναι η σύστασή σας προς τον διάδοχό σας ώστε να μειωθεί αυτή η τόσο μεγάλη διαφορά. Πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τις δυνατότητες που έχουμε, τις τεχνικές, τις, χρηματο... τις οικονομικές, αλλά και του ανθρώπινου μας δυναμικού για να μπορέσουμε να ε, αναπτυχθούμε κατά τέτοιο τρόπο και να συμβάλλουμε όσο μπορούμε ε, και εμείς στην ε, Ευρώπη. Ποια θα είναι η σύστασή σας λοιπόν για να μειωθούν οι διαφορές μεταξύ παλαιών και νέων κρατών μελών. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Now the last coordinator will be... Σας ευχαριστώ κύριε Τουζανόφσκι. Τελευταία συντονίστρια κυρία Βέρα από την ΚΟΕ, σας ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό και η ανάπτυξη τεχνολογική και η ανάπτυξη αρμοδιοτήτων και η συνεργασία με τις άλλες χώρες καθώς και η ειδίκευση. Γι' αυτό θεωρούμε πως η συμβολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας όπως και άλλες μορφές ε, χρήσης του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού μπορεί να συμβάλλουν ε, σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη την οικονομική και την κοινωνική στην Ευρώπη καθώς προωθούν καλύτερη ποιότητα ζωής και πολιτικές ε, για όλους. Η ανάλυση που κάναμε για την αποστολή και την αξιολόγηση της ε, τυπολογίας των υποτροφιών που έχουν δοθεί δημιουργεί όμως ερωτήσεις. Ε, πρώτον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας έχει κάποιο ε, είδος κριτηρίου όπως η αποκέντρωση για την χορήγηση των ε, υποτροφιών. Ας πούμε, το 2019 χρηματοδοτήθηκαν 408 προγράμματα. 57% αυτών των προγραμμάτων αφορούσε τέσσερις χώρες. Γερμανία 18%, Γαλλία 10%, η Ολλανδία 13% και Ηνωμένο Βασίλειο ε, άλλο ένα 10%. Η Πορτογαλία έλαβε χρηματοδότηση για δύο προγράμματα που συμβάλλουν στην δημιουργία έρευνας τα νούμερα δείχνουν ότι περισσότερο ε, σε αιτήσει υποβάλλουν αυτές οι χώρες ή ότι δεν υπάρχουν κριτήρια που να ενισχύουν ε, την ε, συνοχή σε εδαφικό επίπεδο. Έπειτα, οι υποτροφίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας σημαίνουν ε, ε, τη ε, σύναψεις συμβάσεων με σεβασμό στις ε, συνθήκες απασχόλησης, ώστε δηλαδή να υπάρχουν εγγυήσεις ότι τα χρήματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας δεν χρηματοδοτούν ε, επισφαλείς θέσεις απασχόλησης, αλλά συμβάλλουν στην ε, ανάπτυξη, στην επιστημονική έρευνα και κατά τη γνώμη μας το μέλλον χρειάζονται αυτές οι σταθερές συνθήκες εργασίας έπειτα η στατικοποίηση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει ότι θα πρέπει να ε, ελεγχθούν από στρατιωτικής αξίας τα project τα οποία χρηματοδοτούνται. Ποιο ποσοστό της χρηματοδότησης πάει σε τέτοιου φύσεις project. Ευχαριστώ. Thank Now we have Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τώρα ακόμα πέντε συναδέλφους που θέλουν το λόγο, οπότε παρακαλώ να έχετε υπόψη ότι στι 12.30 τελειώνει η συνεδρίασή μας. Παρακαλώ. Εγώ θέλω να ξεκινήσω με μια δήλωση. Το ΕΛΚΑ θα στηρίξει την ανεξαρτησία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνα με κάθε τίμημα και με κάθε μέσο. Πρόκειται για ένα θέσμα για την αριστεία, για την ε, σύγκριση των νομοτήμων. Έχουμε επίσης τα κράτη-μέλη και δεν υπάρχει ελευθερία της έρευνας à la carte. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες ε, όσον αφορά τη γεωγραφική ισορροπία για τα θέματα κλιματικών αλλαγών, αλλά δεν μπορεί το ERC είτε είναι ανεξάρτητο, αλλά να είναι ανεξάρτητο να λέμε ναι, αλλά το 35% θα πρέπει να πάει για τις κλιματικές αλλαγές και την ισορροπία των φύλων και τη γεωγραφική ισορροπία κτλ. Τότε δεν θα είναι πια το ERC, ε, γιατί αυτό πρέπει πρέπει να έχει να κάνει με την αριστεία. Διαφορετικά δεν ισχύει πια το πράγμα. υπάρχουν πτυχές όπου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, αλλά πάντως δεν θέλουμε εμείς να πλήξουμε την εξαρτησία του ERC. θα χρησιμοποιηθεί αυτό ως κριτήριο για να γράψουν την ατζέντα του ERC. Εμεί δεν επιθυμούμε να το κάνουμε αυτό, αν και θεωρούμε πως είναι σημαντική η πτυχή, αλλά δεν εφαρμόζεται από άλλους, από την Κομισιόν, το Κοινοβούλιο κτλ. Το ERC πρέπει να είναι ανεξάρτητο, γιατί διαφορετικά η σημασία αυτής της παγκόσμιας διάστασης του ERC είναι ακριβώς η ανεξαρτησία του οργανισμού αυτού που βασίζεται στην εξέταση των ομοτήμων, στην αριστεία. Θα το καταστρέψουμε αυτό και θα είναι απλά άλλο ένα κομμάτι ενός οποιοδήποτε προγράμματος. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι και για τα θέματα φιλοδοξίας και ερωτήσεων για τη γεωγραφική ισορροπία, ναι, ρωτήστε αλλά δεν θα πρέπει να ε, σημαίνει οποιοδήποτε περιορισμό στην ελευθερία του ERC, γιατί διαφορετικά το διαλύουμε αυτό το μέσο και αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβουμε. Η ερώτησή μου είναι τι θα γίνει, μιλήσαμε για περισσότερα χρήματα, αλλά ήδη σήμερα το πρωί συναντηθήκαμε με την Κομισιόν και το Συμβούλιο θα αποφασίσει για μια κοινή θέση υπό την Φιλανδική Προεδρία, αλλά μιλάμε για περικοπές 12 δις Ερώτησή μου είναι, εσείς ασκείτε πίεση με τον παραδοσιακό τρόπο των ευρωπαϊκών θεσμών. Το ERC δεν θα έπρεπε λίγο περισσότερο να επιμείνει, γιατί αν περικοπούν αυτά τα 12 δις, μιλάμε για περικοπή μεγάλη. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν ώστε να δημοσιοποιηθεί αυτή η υπόθεση, ότι δηλαδή αν μειωθούν 12 δις αμέσως σημαίνει περικοπή 2-3 ε, δις για το ERC και άρα περικοπή των φιλοδοξιών του οργανισμού. Η κυρία Τόγια. Ε, ναι, ευχαριστώ. Και εγώ θέλω, όπως και οι συνάδελφοί μου, να ευχαριστήσω τον κύριο Μπουργκινιόν για την εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει και που έχει δείξει και έχει προωθήσει την αριστεία προς όφελος όλων των χωρών της Ένωσης. Εγώ προσωπικά είδα τη χώρα μου να, στη χώρα μου να αναπτύσσεται η προσοχή και η δυνατότητα επαφή και αλληλεπίδραση με τον οργανισμό αυτό. Ευχαριστούμε λοιπόν. Η δεύτερη μου παρατήρηση είναι κάτι που είπαν όλοι οι συνάδελφοι, ότι εμείς υπερασπίζουμε αυτή την πραγματικότητα, την υπερασπίζουμε στο ορίζον, όπως υπερασπίζουμε ολόκληρο το πακέτο και νομίζω πως ο καθένας θα πρέπει να ε, κάνει τη φωνή του ακούστη, Να έχουμε δηλαδή στον ερευνητικό κόσμο με τα στοιχεία στα χέρια μας ε, να στηρίξουμε ότι πρέπει αυτόν τον οργανισμό. Νομίζω όμως βασικό έργο είναι των πολιτικών. Εμείς πρέπει να καταλάβουμε τι δουλειά θέλουμε να κάνουμε και να ε, συμβάλλουμε στην στήριξη αυτού του οργανισμού. Τώρα, αυτή ο φόβο που έχει δημιουργηθεί με την προετοιμασία του Horizon ε, Europe ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό ε, Ερευνητικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Κοινοτομία δεν θα πρέπει να υπάρχει. Γιατί και οι δύο πυλώνες είναι σημαντικοί. Ο νέος πυλώνας δεν θα πρέπει να αποδυναμώσει το ERC. Μάλιστα πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο και έχω και προτάσεις ε, που να είναι πιο συμπληρωματικά αυτά τα δύο τόσο σημαντικά στοιχεία. Είναι διαφορετικά τα πλαίσια, αλλά δεν είναι διαφορετικός ο κόσμος, είναι ο ίδιος κόσμος, ο ευρωπαϊκός. Οπότε, για την ανεξαρτησία του πρώτου και την ανεξαρτησία του δεύτερου να δημιουργηθούν ε, δυνατότητες συνεργασίας. Ε, μια πιο ολοκληρωμένη λοιπόν έρευνα χωρίς να χάνουμε τις ιδιαιτερότητες. Και τελευταία παρατήρηση πιστεύω και εγώ ότι πρέπει να βρούμε μέσα Κάθε περίοδος έχει τις προτεραιότητές της. Να βρούμε μέσα, να επιβεβαιώσουμε τις προτεραιότητες του ERC, την μακροχρόνια έρευνα, τα όσα είπατε εσείς. Πιστεύω πως πρέπει να βρούμε τρόπο να το καταστήσουμε πιο, όπως έλεγε και η κυρία Καρβάλιο, πιο, πώς να το πω, πιο αξιοποιήσιμο, δηλαδή να, να δημιουργηθεί προσθεθέμενη αξία. οι επιστήμονες βοηθούνται στη δική τους ε, σταδιοδρομία μέσω του ECR. Πρέπει να βρεθούν τρόποι δηλαδή συνεργασίας, να βρεθεί αυτό το πνεύμα, το κοινό, ώστε τα πορίσματα να ε, αξιοποιηθούν περισσότερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. πολύ. Από το Renew. Ο κύριος ε, Πεκαρίνεν. Ευχαριστώ πολύ. Αρχικά θα ήθελα να συμφωνήσω με τα όσα είπε ο κύριος Έρες. Η αριστεία. θα πρέπει να είναι το πιο σημαντικό κριτήριο. Είναι το μόνο σημαντικό κριτήριο όταν ε, μιλάμε για καινοτομία ε, και για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας. Και θα ήθελα επίσης ε, να συγχαρώ τους εκπροσώπους του Συμβουλίου Ελπίζω επίσης ε, αν ε, θα μπορούσατε να δώσετε κάποια κίνητρα στα κράτη-μέλη, διότι πιστεύω ότι θα πρέπει και τα ίδια να επενδύσουν ε, περισσότερο στην έρευνα και την ε, καινοτομία. Γνωρίζουμε ότι Μονάχα δύο χώρες έχουν καταφέρει να πετύχουν τον ε, στόχο. Χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις ε, στα κράτη-μέλη. Τώρα όμως ε, το ερώτημα είναι ποια είναι η δική σας άποψη. Πώς καλά λειτουργεί η αλυσίδα της ε, καινοτομίας ε, στην Ευρώπη το πώς ε, υπάρχουν δυνατότητες για την καινοτομία, το πώς τις εμπορευόμαστε και το πώς τις παράγουμε σε σύγκριση για παράδειγμα με την Νότιο Κορέα, τις Ηνωμένε Πολιτείε και άλλες χώρες πιστεύω ότι δεν έχουμε προχωρήσει και επιτύχει τόσο πολύ όσο απαιτείται. Ευχαριστώ πολύ και τώρα από τους σοσιαλδημοκράτες η κυρία Μούνιος. Ευχαριστώ πολύ. Ε, συγχαρητήρια για το success stories, όχι, success story, όχι μονάχα ε, για τον ε, τομέα της έρευνας εχμής, αλλά ταυτόχρονα βοηθάει και στην ε, προώθηση των εθνικών δομών έρευνας σε διάφορες χώρες. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, είναι ξεκάθαρη επιρροή η ελευθερία και η ε, ανεξαρτησία την οποία είχατε πιστεύω ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ε, ρόλο. Ισχύει ε, ότι θα πρέπει να προωθήσουμε και τις δυνατότητες ε, και για τις ε, περιοχές όπου δεν υπάρχει μεγάλη προσώπηση στον τομέα της έρευνας. Ε, πώς λοιπόν πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις τόσο όσον αφορά τον διαμοιρασμό των, της χρηματοδότησης σε αυτές τις περιοχές αλλά και το πώς θα μπορέσουμε να προωθήσουμε την ισότητα ε, των φίλων όσον αφορά την ε, χρηματοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Και η κυρία Καηλή από τους Σοσιαλδημοκράτες. Uh, ε, γνωρίζω πόσο ενεργός ήσασταν, κύριε καθηγητά σε πολλούς τομείς ε, και το πόσο σημαντικό είναι να ε, κατανοούμε την αριστεία για να μπορέσουμε να προωθήσουμε ένα τόσο σημαντικό έργο και πιστεύω ότι ε, είναι σημαντικό να γίνουμε ανταγωνιστικοί σε σχέση με τη ΣΥΠΑ και, της, και την Νότιο Κορέα. Δεν ήταν κάτι εύκολο αυτό. Έχει υποθεί επανειλημμένο σε αυτό και εφόσον προσπαθούμε να προωθήσουμε και να παρουσιάσουμε όλα τα επιτεύγματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, θα ήθελα ε, να ρωτήσω εάν υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε ούτως ώστε να προωθήσουμε τη διασυνοριακή συνεργασία και ε, έτσι να συμμετάσχουν και τα ε, κράτη-μέλη ε, τα οποία ίσως να μην ξέρουν για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνα. Γνωρίζω ότι η αριστεία προσελκύει η αριστεία, όμως ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα ούτως ώστε περισσότεροι ερευνητές, επιστήμονες και πανεπιστήμια να συμμετέχουν και να συνεισφέρουν. Οπότε έχουμε τη διασυνοριακή έρευνα και επίσης αν έχετε κάποια άποψη σχετικά με το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια υποχρέωση ούτω ώστε να επιστρέφουν κάτι αυτοί οι οποίοι επωφελούνται από αυτήν την έρευνα. Δεν εννοώ γενικά, αλλά συγκεκριμένα ε, στον τομέα της ανάπτυξης, πατέντες, ε, ε, IP, πνευματική ιδιοκτησία. Ε, πώς όλα αυτά μπορούν να ε, χρησιμοποιηθούν. Ε, αυτό θα βοηθούσε ούτως ώστε το Συμβούλιο Έρευνας να είναι πιο δυνατό κάθε χρόνο. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Καηλή και τώρα η κυρία Σολής Πέρες. Ευχαριστώ κυρία Μπουργκινιό. Θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η άποψή σας για αυτό στο οποίο αναφέρθηκε νωρίτερα. Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε τις δραστηριότητες καινοτομίας στα πλαίσια του ERC και τα project που χρηματοδοτούνται από το ERC ε, ε, θα πρέπει να έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία και στην οικονομία. Και υπάρχει ένα εργαλείο, ένα ειδικό εργαλείο, το Proof of Concept, το οποίο λειτουργεί πολύ καλά. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψή σα για το κατά πόσο πρέπει να δοθούν μεγαλύτερα κονδύλια στα προγράμματα όπως το Proof of Concept ή αν πρέπει να επικεντρωθούμε στην βασική έρευνα ε, που επίσης υποχρηματοδοτείται. Το δεύτερο ερώτημά μου έχει να κάνει με αυτή την Ευρώπη των δύο ταχυτήτων στην έρευνα. Υπάρχει ισορροπία μεταξύ των χωρών. Ε, τι θα πρέπει να κάνουμε για να συνεισφέρουμε έτσι ώστε αυτή η ισορροπία να αποκατασταθεί. Ευχαριστώ. So much. Now. Ευχαριστώ πολύ. Αρκετές οι ερωτήσεις και οι παρεμβάσεις. Παρακαλώ. Κύριε ε, Μπογιόν και κύριε Ε, έχουμε ερωτήσεις ε, οι ε, όπως είναι για παράδειγμα της κυρίας Καβάλιου, το Συμβούλιο Αρεύνας λοιπόν ε, έχει κάνει έτοιμα ε, ε, σχετικά με το πλαίσιο του, σχετικά με το πι. θεωρούμε ότι η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για το Συμβούλιο Έρευνας, το προσωπικό εκεί μπορεί να συλλέξει και να οργανώσει τα αποτελέσματα της έρευνας πρόκειται για, για έναν εκτελεστικό οργανισμό, δεν είναι κομμάτι της αποστολής του και πιστεύουμε ότι, ότι το να έχουμε μια παγκόσμια εικόνα των αποτελεσμάτων είναι μια ευθύνη που θα πρέπει να ε, δοθεί. Και σίγουρα ο ρόλος του ERC δεν είναι ε, να νομοθετεί ε, Σίγουρα όμως αυτοί οι οποίοι παρακολουθούν ε, την ε, βελτίωση του προγράμματος ε, μπορούν να κρίνουν καλύτερα γι' αυτό. Είναι μια ένα ξεκάθαρο αίτημα το οποίο θέσαμε. Αναφέρεται στο Horizon 2020 ότι θα συμβεί και ίσως το Κοινοβούλιο θα μπορέσει να βοηθήσει πάνω σε αυτό. Το επόμενο θέμα τώρα σχετικά με το πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τις δραστηριότητες του ERC με άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο του Horizon 2020 αναφέρθηκε από ε, κάποιους ε, ευρωβουλευτές φυσικά και δεν περιμέναμε ότι αυτό ε, υπάρχει για να μπορέσουμε να ε, εργαστούμε πάνω σε αυτό. Εμείς ε, καλέσαμε τα μέλη της ομάδας υψηλού επίπεδου για να συζητήσουμε πάνω σε αυτό, να τους παρουσιάσουμε το πώς εργαζόμαστε, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε γέφυρες συνεργασίας και ήδη έχουμε κάποιες συζητήσεις με τον κύριο ε, που είναι υπεύθυνο ε, για την ε, δημιουργία της Task Force για το Συμβουλίο Έρευνας. Δεν θα είμαι όμως εκεί, διότι η εντολή μου, η θητεία μου μάλλον τελειώνει τον Δεκέμβριο. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερο κάτι το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί έχουμε το πλαίσιο ε, απόδειξης ε, σχεδίου το οποίο ε, θα προωθηθεί, το οποίο σημαίνει ότι κάποια από τα προγράμματα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί από το ERC, ότι είναι προγράμματα τα οποία έχουν περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης, θα πρέπει να τα προχωρήσουμε σε άλλο επίπεδο τώρα. και θα πρέπει φυσικά να υπάρξει η δυνατότητα χρηματοδότησης. Ε, ε όμως αυτός δεν είναι δικός μας ε, τομέας. Ε, τώρα ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Έχουμε αναπτύξει σχέσεις με το IBAN, θεώρησαν ότι κάποια από τα προγράμματα που έχουμε θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν και έτσι λοιπόν η ιδέα ε, των ερευνητών που έχουν ε, ταυτοποιηθεί για αυτό δεν ανταποκρίνεται τόσο στην ε, πραγματικότητα. Το Horizon Europe θα πρέπει να ε, συμβάλλει σε αυτή τη διαδικασία περισσότερο και αυτός θα είναι ένας ε, τρόπος με τον οποίο το ERC θα μπορέσει να συνεισφέρει περισσότερο. Θα πρέπει βέβαια να σεμβόμαστε την ε, αρχή του από κάτω προς τα πάνω και αν δεν το κάνουμε αυτό τότε θα έχουμε προβλήματα. Τώρα όσον αφορά την δημοσιοποίηση, κάτι το οποίο ανέφερε ο κύριος Νίκα. Έχουμε κάνει ε, προσπάθειες ούτως ώστε να γίνει πιο ορατό το ERC. Είχαμε δράσει στο Κοινοβούλιο με την κυρία Στόα, είχαμε εκδηλώσεις δύο φορές ε, στο Κοινοβούλιο. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν ε, τόσα πολλά ε, προγράμματα της Επιτροπής για την έρευνα που να παρουσιάζονται τόσο πολύ στο Κοινοβούλιο ο πρόεδρος του ε, Κοινοβουλίου μας έκανε την ε, τιμή να παρευρεθεί. Έχουμε κάνει, ε, έχουμε, κάνουμε μεγάλη προσπάθεια στον τομέα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. λαμβάνουμε υποστήριξη από τους επιστήμονες που υποστηρίζουμε και από την Επιτροπή. Ε, και επίσης έχουμε τα ERC Comics όπου συνεργαζόμαστε με καλλιτέχνες ε, που ε, σχεδιάζουν κόμικ και με ερευνητές και η επιτυχία είναι ότι οι ερευνητές και οι καλλιτέχνες συνεχίζουν και συνεργάζονται μετά το πρόγραμμα αυτό. Έχουμε κόμικ online όμως σκεφτόμαστε επίσης να τα τυπώσουμε κιόλας σε αυτούς ε, τους τομείς λοιπόν είμαστε πραγματικά αποφασισμένοι ε, και πιστεύω ότι και ο διαδοχός μου θα ε, συνεχίσει να κάνει παρόμοιες προσπάθειες. Τώρα όσον αφορά το θέμα της κοινή συνεργασίας με τα κράτη-μέλη ήταν ένα θέμα το οποίο με αποσχόλησε Ε, μιλάμε για διαφορετικές δομές, διότι κάθε κράτος μέλος είναι διαφορετικά οργανωμένο. Αυτό το οποίο προωθούμε λοιπόν είναι σε τοπικό επίπεδο διάφορες ε, εθνικές ε, υπηρεσίες ή διάφοροι ιδιωτικοί οργανισμοί σε τοπικό επίπεδο λοιπόν ε, ε, όσους έχουμε επιλέξει από το Συμβούλιο να λάβουν μια ε, χρηματοδότηση να τους δώσουμε τη δυνατότητα που έχουν επιλογή ως άριστοι από το Συμβούλιο Έρευνας αλλά δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση να βοηθηθούν σε εθνικό επίπεδο. Εδώ λοιπόν είναι ένας τομέας όπου θα μπορούσαμε να δούμε μια περαιτέρω συνεργασία με τα διαρθρωτικά ταμεία. Το έχουμε προσπαθήσει, δεν έχει προχωρήσει αρκετά. Δηλαδή, διότι ο κανονάς ε, σχετικά με τη χρήση των διορθωτικών ταμείων είναι ξεκάθαρος ε, οπότε ε, δεν υπάρχει τόση ευελιξία εδώ πέρα. Να είναι λοιπόν κάτι σημαντικό για τα προγράμματα του ERC. οι διαφορετικές ε, συνθήκες υποστόρεξης ε, έρευνας ε, στα κράτη-μέλη είναι αξιοσημείωτη. Σε, κάποιος, σε δύο κράτη-μέλη είναι πάνω από το 3% και υπάρχουν από την άλλη χώρες στην έρευνα όπου υποστήριξη, υπάρχουν άλλες χώρες όπου η υποστήριξη στην έρευνα είναι κάτω από το 0,5%. Και φυσικά λοιπόν δεν θα πρέπει να τιμωρηθούν ε, αυτές οι χώρες επειδή δεν έχουν πρόσβαση σε πόρους, αλλά θα πρέπει να υπάρχει βοήθεια. Εν τέλει όμως ε, δημιουργείται ε, μία ανισότητα Δυστυχώς όμως αν αλλάξουμε τα κριτήρια ε, και είναι αποκλειστικά η επιστημονική αριστεία, τότε ε, πολύ ε, πιθανόν κάποιοι να μην κάνουν αίτηση και επίσης δεν θα μπορούμε να προσελκύουμε τους ερευνητέ για να αξιολογούν τα υπόλοιπα προγράμματα αν θα γνωρίζουν ότι θα πρέπει να κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μας απασχολεί. Με, προσωπικά με απασχολεί πολύ Έχουμε συνεργάτη, για παράδειγμα, στην ε, Ρουμανία. Γνωρίζω ότι έχει πάρα πολλούς πάρα πολύ καλούς μαθηματικούς και εγώ είμαι μαθηματικός και θα πρέπει να ε, διασφαλίσουμε ότι οι τοπικές δομές υποστηρίζουν ε, τους ερευνητές, τους επιστήμονες εκεί ούτως ώστε να έχουν ένα κίνητρο να υποβάλουν την πρότασή τους. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Μποέτιους. Έχω εργαστεί και εγώ σε διάφορα πάνελα για πολύ καιρό και έχω συζητήσει ε, και για στήματα επιστημονικής επικοινωνίας. Υπάρχει μια συζήτηση και μια υποστήριξη σε ό,τι αφορά την άμεση πρόσβαση, στην ανοιχτή πρόσβαση της επικοινωνίας. Είναι μια συζήτηση που γίνεται για να ενισχυθεί αυτή η ανοιχτή πρόσβαση. Όλα τα στοιχεία που προκύπτουν ε, ε, αποτελούν μέρος της επιστημονικής γνώσης και είναι προσβάσιμα σε όλους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, ε, επειδή θεωρείται ε, μια, ένα βραβείο πολύ σημαντικό, θα ζητηθεί από όλου του ανθρώπου, όχι μόνο από τη χώρα του και από το project, αλλά και από τα πανεπιστήμια, να μιλήσουν, να επικοινωνήσουν, να δείξουν ποιε είναι αυτέ οι μεγάλε ιδέε ε, και βεβαίως αυτό ε, προσελκύει και νέους ανθρώπους να κάνουν PhD. Ε, νέα ταλέντα λοιπόν που συνεργάζονται μαζί τους, μην τα ξεχνάμε αυτά, διότι όλα αυτά βασίζονται στην αριστεία. Να σας πω επίσης, επειδή ήμουν σε ένα πάνελ μου τέθηκε ένα ερώτημα για το τι θα άλλαζα. Όταν είναι κάποιος σε ένα πάνελ, επιλέγει από πολλά CV, από πολλές ιδέες. Ε, το πρόβλημα είναι ότι επειδή υπάρχει χαμηλή χρηματοδότηση, ε, όταν ξέρουμε ότι είναι πολύ μεγάλη διαφορά με την υποτροφία ε, και ξέρουμε ότι τα χρήματα δεν ήταν αρκετά ε, για να φτάσει τον επόμενο υποψήφιο από την χή χώρα ή από το χ φύλλο και αυτό πραγματικά είναι οδυνήρο δεν πρέπει λοιπόν να απορρίπτουμε διάφορες ιδέες που είναι A-rated. Ε, τέλος. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποιες χώρες δεν έχουν αρκετές ευκαιρίες. Ε, όταν κάποιος επενδύει στην επιστήμη αυτό έχει αποτέλεσμα, έχει απόδοση. Ε, αυτό που δεν πρέπει να γίνει είναι να μειωθεί ο προπολογισμό, διότι αυτό μειώνει τις πιθανότητες διότι τότε θα επιλέξουμε αυτούς που ούτως ή άλλως έχουν το καλύτερο περιβάλλον να εργαστούν. Είμαι λοιπόν πεπισμένη ότι, ότι το ERC είναι ένα από τα στοιχεία που μπορεί να βοηθήσει, αλλά είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το δούμε αυτό σε σχέση με τις γιγαντιές επενδύσεις που γίνονται από άλλες χώρες και εγώ στη Γερμανία πρέπει να ασχοληθώ με το θέμα των πολιτικών ε, που ακολουθούνται στην Κίνα. Ε, έχουν ένα πρόγραμμα αναζήτησης ταλέντων, ε, τα οποία συχνά τα παίρνουν από την Ευρώπη και τους δίνουν σημαντική ελευθερία, με σημαντική χρηματοδότηση. Γι' αυτό είναι ο τρόπος, μας το δείχνουν άλλες χώρες αυτά. Ήθελα να αναφέρω Το ERC είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα για την καινοτομία μας, για την έρευνά μας. Γνωρίζουμε, γνωρίζουμε από την ιστορία των επιστημών ότι η καινοτομία και η όπως και η αριστεία δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να κάνει προγραμματίσει ε, αλλά χρειάζεται υπομονή ε, και χρειάζεται και διάδραση συχνά ζητώνται ζητείται από τους ερευνητές, από τους πολιτικούς, από τα, τις επιχειρήσεις, ε, ε, από, από τα πανεπιστήμια να κάνουν μια προσπάθεια να επικοινωνήσουν περισσότερο και δεν πρέπει να το αποτιμήσουμε αυτό. Ε, Σας ναι. ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μπουργκίνο, ναι, δύο ακόμα παρατηρήσεις. Η μία είναι ο αριθμός των χωρών που έχουν πραγματικά εισάγει μεταρρυθμίσεις στο ερευνητικό του σύστημα. Το πιο εντυπωσιακό παράδειγμα είναι η Πολωνία που δημιούργησε το NCN που είναι ε, το βασικό έδημα και η μεταρρύθμιση των πανεπιστημίων που μόλις έγινε και τους δίνει περισσότερες δυνατότητες να αναπτύξουν έρευνα σε υψηλό επίπεδο. Δεύτερη παρατήρηση για το ερωτικό σα ερώτημα που αφορά την υποχρέωση, τη φιλόδοξη μάλλον, τη φιλοδοξία για να έχουμε περισσότερους πόρους για τις κλιματικές αλλαγές. Αυτό το οποίο δεν βρίσκω θετικό είναι όχι η προτεραιότητα αυτή καθ' αυτή, Βλέπετε, φορώ και εγώ αυτή την κονκάρδα που σημαίνει μια δεσμεύση πολύ σημαντική, αλλά η δυσκολία είναι να μετράμε κάθε φορά τα χρήματα. Εμείς πρέπει να συνδυάσουμε την αξιολόγηση και της ποιότητας, γιατί ξέρετε ότι ανάμεσα στα προγράμματα, και αυτό το έχω κάνει πολύ συστηματικά για την, ε, για την ε, ε, ενέργεια, ξέρετε ότι ορισμένα project αλλάζουν τελείως τα τοπία και ακόμα αν τα ποσά που πήγαν εκεί δεν ήταν τόσο σημαντικά, ο τελικός αντίκτυπος ήταν πολύ μεγάλος. Σε άλλες περιπτώσεις υπάρχει μια μακρά και σταθερά προσπάθεια που όμως δεν θα αλλάξει τίποτα γρήγορα. Για μένα λοιπόν η δέσμευση για το περιβάλλον, για τις κλιματικές αλλαγές θα πρέπει να έχει δύο διαστάσεις. Η μία είναι σημαντική προσπάθεια, ναι, αλλά όσον αφορά τα ποσοστά και τα χρήματα, αλλά ταυτόχρονα να εντοπίσουμε ποιες είναι οι προτάσεις, τα project, νέες ε, δηλαδή εξελίξεις ε, που αλλάζουν τελείως τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα. Και ε, είδαμε και πολύ καλό παράδειγμα στη δική σας εργασία, ότι δηλαδή υπάρχουν πράγματα που μπορεί να αγνοούσαμε τελείως ή να παρερμηνεύουμε. Και τελικά να μην αντιμετωπίζουμε το θέμα. Ας πούμε, όσον αφορά την ε, τήξη του, των πολικών παγετώνων, ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε. Και βλέπουμε πως ε, ε, λιώνει ο πολικός παγετώνος πολύ πιο γρήγορα από ότι πιστεύαμε και η, η, η σχετική έρευνα ήταν πολύ σημαντική για να μπορέσουμε να κάνουμε τις σωστές μετρήσεις. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο το χρήμα που μετράει, είναι το θέμα και η ποιότητα της ε, ε, έρευνας και το αντικτύπου αυτής. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βουργινιό και κυρία Μποετίους που ήρθατε και μοιραστήκατε μαζί μας τις προπτικές και τους προβληματισμούς σας. Πολύ ενδιαφέροντα ήταν όλα αυτά και έτσι κλείνουμε την πρωινή μας συνεδρίαση και θα ξαναρχίσουμε στις 2.30. Σας ευχαριστώ.